Παρακαλώ, συνάδελφοι, καθίστε. Πρέπει να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα πολύ σημαντικό σημείο στην ημερήσια διάταξη, ανταλλαγή απόψεων με την Επίτροπο Βασιλείο για την ε, οδηγία για, τα, ε, για τις παροχές υγείας ε, διαμεθοριακά σε ασθενείς. Καταρχάς να καλωσορίσω την κυρία Βασιλείου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι θα ανταλλάξουμε απόψεις για το θέμα αυτό, διότι η Επιτροπή μας συμμετείχε ενεργά στο ζήτημα αυτό. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό οι υπηρεσίες υγείας όπως και οι άλλες υπηρεσίες να υποστηρίζονται για τους πολίτες ε, διαμεθοριακά και για τους ασθενείς αφενός και για όσους παρέχουν υπηρεσίες υγείας αφετέρου. Να σας δώσω το λόγο λοιπόν κυρία Βασιλείου. Αξιότιμα μέλη, χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι μαζί σας εδώ σήμερα. Καταρχάς να σας ευχηθώ καλή χρονιά και ό,τι καλύτερο Ξέρω ότι πλησιάζουν οι πολύ σημαντικές εκλογές ε, και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο στην, ε, στις προσπάθειές σας. Το 2009 σαφώς θα είναι μια χρονιά αλλαγών και προκλήσεων για όλους μας και ελπίζω και ότι θα είναι και μια χρονιά επιτυχίας και καλής υγείας. Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για μένα να συζητήσω μία από τις σημαντικότερες οδηγίες στον τομέα της υγείας την οποία έχει ε, θέσει ως προτεραιότητα, έχει παρουσιάσει η παρούσα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρόταση για την οδηγία για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών σε παροχές ε, υγείας διαμεθοριακά. Ξέρετε πάρα πολύ καλύτερα από μένα ότι όταν ε, η υγεία αποκλείστηκε από την Οδηγία για τις Υπηρεσίες το 2006, εσείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητήσατε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ετοιμάσει μια συγκεκριμένη πρόταση που θα λάβει υπόψη τις ιδιαιτερότητες και την περιπλοκότητα του τομέα της υγείας. Το κείμενο της πρότασης ε, προέκυψε ως αποτέλεσμα μιας δημόσιας διαβούλευσης που ξεκίνησε το 2006 μια αξιολόγηση αντικτύπου και μια έρευνα του, του Ευρωβαρομέτρου που έγινε το 2007 και επίση του έργου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κινητικότητα των ασθενών και τι υπηρεσίε υγεία. Αναφέρομαι στι εκθέσει του κυρίου Μπόη από το 2005 και τη κυρία Βερνιόν από το Μάιο του 2007. Η πρότασή μας ουσιαστικά αντικατοπτρίζει τι ιδέε και τι αρχέ που παρουσίασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτέ τι πολύ σημαντικέ εκθέσει. Δεν θα επισέλθω σε όλες τις λεπτομέρειες αυτής της πρότασης. Είμαι βέβαιη ότι οι περισσότεροι από εσά την έχουν διαβάσει και την έχουν μελετήσει ιδιαίτερα προσεκτικά, αλλά θα ήθελα να σα επισημάνω τα βασικά τη στοιχεία. Ο βασικό τη στόχο είναι να δώσει στους ασθενείς καλύτερε ευκαιρίε και πρόσβαση σε υπηρεσίε υγεία ανά την Ευρώπη διότι οι ασθενείς βρίσκονται στο επίκεντρο αυτού του σχεδίου νομοθεσίας. Εκείνο βέβαια που θα πρέπει να σας εξηγήσω επίσης είναι ποιος δεν είναι ο στόχος τους. Η πρόταση δεν ασχολείται με θέματα κινητικότητας ε, εργαζομένων ε, υγείας, ούτε ε, με θέματα εγκατάστασης όσων παρέχουν υπηρεσίες υγείας. Αυτά αντιμετωπίζονται ξεχωριστά από την κινητικότητα των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας, διότι αυτά έχουν να κάνουν με το εργατικό δυναμικό σε θέματα υγείας που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον περασμένο Δεκέμβριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια πράσινη βίβλο για το εργατικό δυναμικό για την υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ξεκίνησε μια δημόσια διαβίλευση προκειμένου να αντιμετωπίσουμε όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με το εργατικό δυναμικό σε τομείς υγείας με ε, συνεκτικό και ολιστικό τρόπο. Είμαι βέβαιη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεισφέρει τα μάλα για να καθορίσουμε τα επόμενα σημαντικά θέματα ε, για, τα, ε, για τους ε, επαγγελματίες στον τομέα της υγείας. Να περάσω τώρα στην πρόταση οδηγίας. Εδώ έχουμε τρεις βασικούς στόχους. Καταρχάς θέλουμε να διευκρινίσουμε τις συνθήκες βάσει των οποίων οι ασθενείς θα έχουν δικαίωμα σε διαμαθοριακές υπηρεσίες υγείας και θα έχουν και δικαίωμα αποζημίωση στη χώρα τους εάν αποφασίσουν ότι αυτή είναι η καλύτερη λύση για αυτούς. Δεύτερον, θέλουμε να διώσουμε διασφάλιση ως προς την ποιότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών υγείας ε, σε όλη την Ευρώπη και να έχουμε και καλύτερη συνεργασία μεταξύ των συστημάτων υγείας. Για τον πρώτο στόχο, η πρόταση αυτή αντικατοπτρίζει τις πολλές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών να αναζητούν ε, παροχές υγείας στη χώρα της επιλογής της και να ζητούν αποζημίωση γι' αυτό, ε, σεβόμενοι ταυτόχρονα και τα συστήματα υγείας των κρατών μελών. Αυτή την προσέγγιση την υποστηρίζουν και το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι θα πρέπει να δώσουμε στους ε, πολίτες μας και σαφήνεια και επαρκείς πληροφορίες για το δικαίωμά τους για τις παροχές υγείας. Κατανοώ ότι τους ενδιαφέρουν οι πιθανές επιπτώσεις ε, ε, στα εθνικά συστήματα υγείας και στην βιωσιμότητά τους και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο απασχόλησε ιδιαίτερα την κυρία Βαρνιόν. Θα ήθελα λοιπόν να σας δώσω και κάποιες διευκρινήσεις από αυτού και να σας διασφαλίσω και κάπως. Η αξιολόγηση αντικτύπου έγινε βάσει πολύ σημαντικών στοιχείων από ειδικού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η, των, η κινητικότητα των ασθενών είναι πάρα πολύ περιορισμένη και φτάνει περίπου στο 1% της συνολικής δαπάνης για την υγεία και στο 1% του συνολικού αριθμού των ασθενών κατά πάσα πιθανότητα θα παραμείνει περιορισμένη και αυτό διότι οι περισσότεροι άνθρωποι προτιμούν να θεραπεύονται όσο πιο κοντά στο σπίτι τους γίνεται. Στη Γαλλία, επί παραδείγματι, βάσει των εκτιμήσεών μας, μόνο 100.000 ασθενείς περίπου αποφασίσουν να ζητήσουν θεραπεία σε άλλο κράτος μέλος κάθε χρόνο. Για τη Γερμανία το στοιχείο είναι περίπου 150.000 ασθενείς, για την Πολωνία περίπου 90.000 ασθενείς. Και τα τρία αυτά παραδείγματα βρίσκονται πολύ κάτω από το 1% που σας ανέφερα πριν από λίγο. Η πρόταση λοιπόν δεν έχει στόχο να προάγει την κινητικότητα αυτής αναγνωρίζει ότι το δικαίωμα στην κοινότητα όμως είναι, στην κινητικότητα συγγνώμη, είναι πάρα πολύ σημαντικό για κάποιους ασθενείς ε, που βρίσκονται σε συγκεκριμένες συνθήκες. Οι επιπτώσεις για την ε, ικανότητα των ε, αρχών των υπηρεσιών υγείας για να σχεδιάσουν τέτοια πράγματα λογικά θα πρέπει να είναι αμεληταία. Επιπλέον η πρόταση προβλέπει και έναν αριθμό δικλείδων ασφαλείας για να ε, αποφύγει τυχόν ε, αναπάντεχες επιπτώσεις. Πρώτον, το πακέτο θα ε, καθορίζεται πάρα πολύ καλά στο, στη... στο κράτος μέλος του ασθενούς. Η πρόταση επιτρέπει σε ένα κράτος μέλος να θεσπίσει ένα σύστημα πρώτερης έγκρισης και δεν θα επιτρέπει σε ασθενείς που ε, αναζητούν ε, την καλύτερη ε, τιμή να δέχονται τέτοιες υπηρεσίες υγείας στο εξωτερικό. Επίσης θα πρέπει να έχει να κάνει και με το πώς λαμβάνεται η αποζημίωση. Η αποζημίωση θα δίνεται βάσει της θεραπείας που θα λάμβανε στη χώρα του ούτως ή άλλως και το κράτος μέλος εξακολουθεί να έχει τον έλεγχο για το κόστος της θεραπείας. Επιπλέον, θα πρέπει να έχουμε ε, εθνικού και περιφερειακού κανόνε οι οποίοι θα συνεσχίζουν να εφαρμόζονται και θα παραμείνουν απαράλλαχτοι. Αν ένα κράτο μέλο χρειάζεται, αν συγγνώμη, ασθενή χρειάζεται διαβούλευση από κάποιον γενικό παθολόγο πριν ε, ειδεί κάποιον ειδικό, αυτό ο κανονισμό, αυτό ο μηχανισμό θα παραμείνει ενισχύ και για όσου αναζητούν ε, υπηρεσίε υγεία στο εξωτερικό με την προπόθεση ότι δεν θα υπάρχει διάκριση. Εάν όμω υπάρχει μια απρόβλεπτη αναζήτηση υπηρεσιών υγείας στο εξωτερικό που θα συνεχίσει να παραμένει πρόβλημα, αυτό δεν θα πρέπει να απειλεί την βιωσιμότητα του συστήματος υγείας. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει μία ακόμα δικλίδα ασφαλείας. Η πρόταση επιτρέπει σε ένα κράτος μέλος να θεσπίσει ένα σύστημα πρώτερης έγκρισης για νοσοκομιακή περίθαλψη. Αυτό θα επιτρέπει στο κράτος μέλος να διασφαλίσει το συνολικά, το σύστημά του βάσει και της νομολογίας του δικαστηρίου. Η πρώτερη έγκριση λοιπόν δεν αποκλείεται, αλλά όπως έχουν αποφασίσει οι δικαστές του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, δεν θα πρέπει να θεωρείται κάτι το δεδομένο. Θα είναι μια εξαίρεση η οποία θα είναι για αποκλειστικά για την νοσοκομιακή περιθέλψη και θα εφαρμόζεται με αναλογικό τρόπο. Αυτά είναι ακριβώς αυτά τα οποία χρησιμοποίησε στην ορολογία του το δικαστήριο. Ο ορισμός επίσης της νοσοκομιακής περίθαλψης είναι πάρα πολύ σημαντικός. Οι ασθενείς θα πρέπει να έχουν σαφήνεια και νομική βεβαιότητα. Θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι δεν υπάρχουν ε, διαφορές ανά την Ευρώπη για τον ορισμό αυτό, διότι ιδάλλως θα έχουμε ανισότητες ανά την Ευρώπη για τους ασθενείς και θα έχουμε και περιττές συζητήσεις και διαφωνίες. Γι' αυτό ακριβώς φρονώ ότι η εισαγωγή ενός συστήματος εθνικής εθνικών καταλόγων για να καθορίσουμε ποια είναι η νοσοκομιακή και ποια είναι η εξειδικευμένη ε, περίθαλψη μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση και να είναι αντιπαραγωγική και θα, δεν θα επιτυγχάνεται ο στόχος της οδηγίας. Πρέπει να διασφαλίσουμε λοιπόν ότι το πνεύμα και η ουσία της νομολογίας του δικαστηρίου διατηρούνται, ιδάλλως ε, θα έχουμε αβεβαιότητα και δεν θα επιτύχουμε το στόχο μας που είναι να διαφυλάξουμε τα δικαιώματα των ασθενών. Να περάσω τώρα στο δεύτερο στόχο της οδηγίας, που είναι να δώσουμε στους ασθενείς μηχανισμούς που θα διασφαλίζουν την ποιότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών υγείας. Σαφής πληροφορίας για να δώσουμε τη δυνατότητα να έχουμε ενημερωμένες επιλογές και κατάλληλες θεραπείες και αποζημιώσεις για τα μέτρα αυτά. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν σαφείς κανόνες σε κοινοτικό επίπεδο σχετικά με το πώς αυτές οι απαιτήσει ε, θα μπορούσαν να ε, γίνουν εφαρμοστές ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν δεν υπάρχουν κανόνες, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ποιότητα και ασφάλεια για τους ασθενείς που διασχίζουν τα σύνορα. Στην έκθεση που εγκρίθηκε το 2007, ζητούσαμε μία ένα ασφαλές, ε, υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικό πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών υγείας ε, διαμεθοριακά. Οι πληροφορίες προς τους ασθενούς εξακολουθούν να είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στο σχέδιο γνωμοδότησης που θα συζητήσετε αργότερα. Το άρθρο 5 του σχεδίου οδηγίας έχει μια σειρά από απαιτήσει για το θέμα αυτό και πιο συγκεκριμένα έχει σαφή ε, πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας, τα οποία θα δημοσιεύουν ε, τα κράτη-μέλη και από εκεί και πέρα θα εποπτεύουν την εφαρμογή τους. Με αυτές τις διατάξεις η νέα οδηγία θα προσδώσει πολύ σημαντικό όφελος σε σχέση με την αρχική πρόταση που είχαμε για την, ε, στην οδηγία για τις υπηρεσίες. Χωρίς αυτά, οι υπηρεσίες υγείας θα αντιμετωπίζονται με τον ίδιο ή με χειρότερο τρόπο, όπως και οποιαδήποτε άλλη εμπορική υπηρεσία και αυτό σαφώς είναι κάτι που δεν επιθυμούμε. Γνωρίζω ότι η διάταξη αυτή θα δημιουργήσει δυσκολίες σε αρκετά κράτη-μέλη, αλλά αν αυτό το άρθρο ε, διαγραφεί, θα παραμελήσουμε ουσιαστικά την ίδια τη φύση της περίθαλψης και θα παραμελήσουμε τους ίδιους τους ασθενείς. Και αυτό θα θέλαμε ακριβώς να αποφύγουμε. Ο τρίτος στόχος για να έχουμε καλύτερη και βελτιωμένη συνεργασία σε κάποιους τομείς. Ε, πολλές φορές αυτά ε, επισκιάζονται και από την επιτυχή της νομολογίας του δικαστηρίου. Έχει σημασία για πολλά θέματα και για τις δυνατότητες που έχουμε για ε, την ανάπτυξή τους ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να δούμε πόσο μεγάλες δυνατότητες έχει η πανευρωπαϊκή ε, συνεργασία για την περίθαλψη. Δεν θέλουμε να αυξήσουμε τη γραφειοκρατία, ούτε να επιβάλλουμε μία ενιαία προσέγγιση για όλους. Θέλουμε να εστιάσουμε σε τομείς όπου μπορούμε να αντιμετωπίσουμε βασικές προκλήσεις και να μπορέσουμε να έχουμε συγκριτικές προσεγγίσεις. Τα δικαιώματα των ασθενών, κυρίες και κύριοι, είναι αποτελεσματικά, σαφή και ασφαλή. Ε, θέλουμε να έχουμε συνεργασία και συνέργειες. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας καλύτερα τις νέες τεχνολογίες και θέλουμε να έχουμε και ενισχυμένη συνεργασία. Αυτά όλα αποτελούν τον κινητήριο μοχλό της πρωτοβουλίας μας. Είμαι βέβαιη ότι συμμερίζεστε και εσείς στις φιλοδοξίες μας και είμαι βέβαιη ότι θα έχουμε μια παραγωγική εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησής σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την εισηγήτρια, την κυρία Βερνιόν, για την πολύτιμη συνεισφορά της. Το σχέδιο γνωμοδότησής της μας δίνει μια πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα βάση για συζήτηση και ελπίζω να σας έδωσα κάποιες ε, ε, χρήσιμες εξηγήσει που είμαι βέβαιη ότι θα συνεισφέρω στη συζήτηση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι φυσικά στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήσεις και να έχουμε μια επικοδομητική συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια της νομοδότησης, την συντάκτρια της νομοδότησης, την κυρία Βερνιόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επίτροπε, κυρία Επίτροπε, για όσα μας είπατε. Προκειμένου να καθησυχαστώ, αλλά δεν είμαι πλήρως ήσυχη από όσα είπατε, κατάλαβα ότι έχετε τρει στόχου, του οποίου συμμερίζομαι κι εγώ. Φαντάζομαι όλοι μα να ορίσουμε του όρου κινητικότητα των ασθενών, να του ε, διαβεβαιώσουμε για την ασφάλεια και την ποιότητα τη περίθαλψη, όλοι συμφωνούμε σε αυτό, και να δώσουμε έμφαση στη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Νομίζω ότι αυτού του τρει στόχου όλοι του συμμεριζόμαστε. Και αυτό για το όφελο των Ευρωπαίων πολιτών. Οι υπηρεσίε υγειονομική περίθαλψη θα πρέπει πάντοτε να συμβάλλουν και στην κοινωνική συνοχή, δηλαδή να μην δημιουργούν ανισότητες μεταξύ των πολιτών σε επίπεδο υγείας και βεβαίως την εδαφική συνοχή, κάτι που απουσιάζει σε έναν βαθμό από την οδηγία. Συμμεριζόμαστε λοιπόν αυτούς τους στόχους, όμως δεν συμφωνούμε απολύτως με το δρόμο που θα έπρεπε να ακολουθήσουμε για να επιτύχουμε τους σκοπούς μας. Σε αυτά που μόλις μας είπατε, κάποια πράγματα με ανησύχησαν διότι μιλήσατε για μελέτη αντικτύπου. όντω η κινητικότητα προς το παρόν είναι το 1% του συνόλου των ασθενών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι μικρό το ποσοστό. Ωστόσο, δεν γνωρίζουμε καθόλου τι θα γίνει με την κινητικότητα των ασθενών, ποιε θα είναι οι ανάγκε του σε μερικά χρόνια σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε ένα ιατρικό περιοδικό της Γαλλίας διάβασα έναν αριθμό που μου έκανε πραγματικά να μπω σε σκέψεις. 54% εσείς αναφέρατε 100.000 Γάλλους ασθενείς που πηγαίνουν στο εξωτερικό για υγειονομική περίθαλψη, είναι μικρός ο αριθμός, αλλά 54% των Γάλλων αυτή τη στιγμή λένε ότι είναι πρόθυμοι να πάνε για υγειονομική περίθαλψη εκτός Γαλλίας. Άρα, εάν σε πολλέ χώρε έχουμε παρόμοια αντανακλαστικά και φαντάζομαι ότι αυτό μπορεί να γίνει και στη Γερμανία, μπορεί να γίνει και στη Μεγάλη Βρετανία, γιατί το, το συζήτησα με ομοσπονδίες ασθενών από πολλές χώρες. Τότε μπορεί όντως να οδηγηθούμε σε σοβαρά προβλήματα. Θα πρέπει η οδηγία αυτή λοιπόν να έχει περισσότερες και μεγαλύτερες φιλοδεξίες. Για τους στόχους σαφώς συμφωνούμε, αλλά θα πρέπει να τους αποσαφηνίσουμε και να διακριβώσουμε πολλά πράγματα. Γιατί παραμένει μεγάλο ποσοστό νομικής αβεβαιότητας. Κυρίως νομίζω δεν θα πρέπει και ελπίζω ότι θα το ξεπεράσουμε αυτό. Ελπίζω ότι η οδηγία αυτή δεν θα είναι ένα εργαλείο για να πράγμα τον ε, ιατρικό τουρισμό. Ε, θα περιοριζόταν σε έναν αριθμό μόνο ασθενών και θα δημιουργούσε ένα σύστημα υγείας δύο ταχυτήτων και πολλές ανισότητες μεταξύ των πολιτών. Ελπίζουμε ότι σε μια τεράστια χώρα, όπως φανταζόμαστε μάλλον, βλέπουμε ότι στις ΗΠΑ που είναι μια τεράστια χώρα, αλλάζει το σύστημα υγείας συνεχώς και δημιουργούνται ανισότητε. Σαφώ. Η Ευρώπη όμω εδώ θα πρέπει να παραμείνει ένα παράδειγμα για του υπόλοιπου. Και για τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών. Η πολυπλοκότητα, η ποικιλία, οι ιδιαιτερότητε του κάθε συστήματο υγεία είναι σημαντικέ. Μην ξεχνάμε ότι σε κάποιε χώρε όπω η Γερμανία, η Ισπανία, Υπάρχουν αυτόνομες περιοχές, υπάρχουν κράτη, κρατήδια, όπου η υγειονομική περιθάλψη παρέχεται με διαφορετικό τρόπο. Ακόμη και αν γενικά υπολογίζεται σε ένα κοινό προπολογισμό. Θα πρέπει αυτά να τα λάβουμε υπόψη. Η έρευνα, οι πληροφορίε, οι ιατρικέ πληροφορίε και οι διοικητικέ πληροφορίε. Νομίζω ότι είναι καθοριστική σημασία τα κράτη-μέλη να συνεργάζονται μεταξύ τους και όχι να έχουμε καταλόγους για να ορίζουμε την νοσοκομιακή ή έξω νοσοκομιακή περίθαλψη εδώ χρειάζονται λοιπόν αποσαφηνήσει. Δεν είναι ακόμη σαφή αρκετά η οδηγία. Η νοσοκομιακή περίθαλψη είναι κάτι που θα πρέπει να το μπορούν να το χορηγούν, να το ε, σχεδιάσουν τα κάτι μελη Εγώ κάνει μια προσπάθεια γιατί θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να υπάρχει πρώτερη έγκριση για την παροχή μέσω των ε, κοινωνικών συστημάτων υγείας που είναι πολύ ευαίσθητα σε όλη την Ευρώπη, είναι πολύ ευάλωτα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήσαμε λοιπόν να ακολουθήσουμε και το δικό σας δρόμο αλλά και το δρόμο των δικαιωμάτων των ασθενών κάνοντας διάκριση μεταξύ πρώτερης έγκρισης που για μένα δεν θα πρέπει να είναι εξαίρεση ή παρέκκληση ε, όταν είναι σημαντική η περίθαλψη που χρειάζεται ένα ασθενή, θα πρέπει το σύστημα κοινωνική ασφάλιση να το γνωρίζει και να μπορεί να καλύψει ε, τι ανάγκε αυτέ. Και η διάκριση γίνεται μεταξύ πρώτερη έγκριση και την αίτηση, α πούμε την βεβαίωση που θα επιτρέψει να φύγει ο ασθενή στο εξωτερικό για να λάβει περίθαλψη που δεν είναι τόσο σοβαρή ίσω. Ε, γιατί νομίζω αυτό θα είναι ένα πλεονέκτημα για του ασθενεί. Όταν θα κάνουν τι δηλώσει του οι ασθενεί, ακόμη και αν δεν χρειάζονται έγκριση, μπορεί να υπάρξει μια θηρίδα, ένα γκισέ που θα τον ενημερώνει για όλα του τα δικαιώματα σε σχέση με το, τα δικαιώματά του, τα διοικητικά και τα ιατρικά ώστε να γνωρίζει ότι στη μια ή στην άλλη χώρα η ποιότητα η ασφάλεια της περίθαλψης είναι έτσι ή διαφορετική και να ξέρει και ποια έγγραφα πρέπει να συμπληρώσει ή όχι. Δεν υπάρχουν λοιπόν νέα δικαιώματα για τους, ε, διαφορετικά δικαιώματα για τους ασθενείς. Θα πρέπει να είναι στην καρδιά των, της μεριμνάς μας και να μην υπάρχουν αντιφάσεις. Ε, επίσης, υπάρχει η έννοια της περίθαλψης που πρέπει να διευκρινιστεί. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό και δεν το έχουμε λάβει ακόμη σοβαρά υπόψη, είναι η συνέχιση, εξακολούθηση της περίθαλψης και της ευθύνης σε περίπτωση προσφυγής ή βλάβης. Σε περίπτωση βλάβης ε, μπορεί να έχουμε διαφορετικές υποθέσεις και επίσης διαφορετική εκδίκαση από το ένα δικαστήριο στο άλλο, από τη μια δικαιοδοσία στην άλλη. Και αυτό μας απασχολεί. Επίσης κάτι άλλο που δεν καλύπτεται και μου φαίνεται σοβαρό είναι να έχουμε βέβαια αναγνώριση των συνταγογραφήσεων. Δηλαδή, ένα ασθενή που θα πάει για περίθαλψη σε μια χώρα θα πρέπει να έχει μια συνταγή από την χώρα του που να μπορεί να αναγνωριστεί, από τη χώρα στην οποία έλαβε την περίθαλψη που να αναγνωρίζεται από τη δική του τη χώρα, στα φαρμακεία, λόγου χάρη. Δηλαδή, μπορεί Εμένα μου έτυχε σε διακοπέ να πάω με συνταγή σε μια χώρα και να μην αναγνωριστεί και η συνταγή μου στο φαρμακείο. Δεν είναι τόσο σοβαρό αυτό, αλλά μπορεί να συμβεί και για σοβαρότερε περιπτώσει. Επίση, Ε, είπατε ότι δεν, ε, είπαμε, μάθαμε μάλλον, δεν πρόκειται να συζητηθεί αυτό ακόμη, αλλά σε επίπεδο νομοθεσία και πολιτική είναι σημαντικό επίση να έχουμε μια θεώρηση τη Ευρώπη και ένα όραμα για το τι θα γίνει σε 15-20 χρόνια. Δηλαδή, είμαστε σε μια ήπειρο που γυράσκει. Και γυράσκει καλά διότι έχουμε παροχές ε, υγείας που είναι καλής ποιότητας. Ζούμε λοιπόν περισσότερο, καλύτερα και αναγκαστικά. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε και νέες υπηρεσίες, θα πρέπει να τις σχεδιάσουμε. Δηλαδή τις, ε, την περίθαλψη μακράς διαρκείας θα πρέπει να σχεδιάσουμε, συμπεριλαμβανομένης της περίθαλψης για τους ε, ηλικιωμένους κατοίκων αυτό νομίζω ότι είναι μια ιδέα πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί θα πρέπει να προστατεύσουμε καλύτερα τους πολίτες και να προλάβουμε τα προβλήματα που σίγουρα θα προκύψουν τα, επόμενα χρόνια. Θα πρέπει λοιπόν και αυτό να το συζητήσουμε νομίζω, να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε το κείμενο και έπειτα. Μια άλλη έλλειψη που μου φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντική δεν γίνεται ιδιαίτερο λόγο για την κινητικότητα των ασθενών, για την ασφάλειά του, για την ποιότητα τη της ε, περίθαλψη σε συνδυασμό με την επαγγελματική κινητικότητα. Δηλαδή, ο συσχετισμό μεταξύ ασθενών και ειδικών των επαγγελματιών του τομέα τη υγεία, δηλαδή των γιατρών, των ε, θεραπών των ιατρών, των νοσοκόμων και το καθεξής, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική. Η οδηγία του 2005 για τα επαγγελματικά προσόντα των ε, επαγγελματιών δεν αρκεί εδώ για να μας καλύψει για, το ιατρικό, για τον ιατρικό κλάδο. Είναι σημαντικό λοιπόν να το λάβουμε και αυτό υπόψη στην οδηγία. Διότι από τη μια έχουμε να κάνουμε με την ποιότητα, από την άλλη με την ασφάλεια, αλλά επιπλέον θα πρέπει να μην το ξεχνάμε ότι ή μπορεί να υπάρξει έλλειψη ισορροπία στην ιατρική δημογραφία, αν θέλετε, στα διάφορα κράτη-μέλη και αυτό ήδη συμβαίνει σε κάποιε χώρε. Άρα μπορει να υπαρξει ελλειψη ισορροπια στην ιατρικη δημογραφια αν θελετε στα διαφορα κρατη μελη και αυτο ηδη συμβαινει σε κάποιες χώρες. αρα η υγεια του πληθυσμού είναι και αυτό μια, ένα εργαλείο για την οικονομική ανάπτυξη σε κάθε περίπτωση, αλλά θα πρέπει να κρατήσουμε και το κοινωνικό μα πρότυπο, το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο. Θα πρέπει λοιπόν να αφιερώσουμε χρόνο σε αυτέ τι ιδέε. Ξέρω ότι πρέπει να προχωρήσουμε και γρήγορα. Είπατε ότι η προτεραιότητα αυτή είναι από τι υψηλότερε για εσά. Είναι πολύ σημαντικό το κείμενο αυτό. Θα υπάρξουν και άλλε για τι υπηρεσίε και το καθεξή. Αλλά είναι πολύ σημαντικό το κείμενο αυτό, αυτή η οδηγία για τη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Βρισκόμαστε σε ένα διάστημα καθοριστική σημασία, κρίσιμο. Α, θα έλεγα ότι περνάμε στη δεύτερη φάση. Θέλουμε να φτιάξουμε οικονομική, κοινωνική και πολιτική Ευρώπη και σημαντικό είναι να μην σφάλουμε, να αφιερώσουμε χρόνο σε αυτά τα θέματα, να τα συζητήσουμε ενδελεχώς και να πάμε στην ουσία των πραγμάτων. Ευχαριστώ, κυρία Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον σκιώδη εισηγητή. Παρακαλώ όμως ε, να μην υπερβείτε τα τέσσερα λεπτά. Ο κύριος Πουπέρκ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο για την παρουσίαση τη σήμερα το πρωί και για τη δουλειά που έχει κάνει μέχρι στιγμής ε, Το σημαντικό με τις υπηρεσίε υγεία είναι ότι είναι ε, πολύπλοκο ε, θέμα, ε, ιδιαίτερη διασυνοριακή ε, περίθαλψη. Δεν είναι κάτι που μπορεί να λυθεί εν μία νυχτή. Νομίζω ότι το σχέδιο που έχει υποβληθεί ε, σε μεγάλο βαθμό παρέχει την απαραίτητη ισορροπία. Τα θέματα που προκύπτουν είναι θέματα όπως είναι οι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, για παράδειγμα στη δική μου χώρα, για συγκεκριμένου τύπου θεραπείες. Ξέρω ότι δεν είναι κάτι στο οποίο μπορεί να υπάρξει ε, διασυνοριακή περίθαλψη, αλλά ε, θα αναγκάσει νομίζω η πρόταση αυτή, ε, θα αναγκάσει τις κυβερνήσεις να κάνουν κάτι. Μια 14χρονη στη χώρα μου πρέπει να περιμένει 5 χρόνια για την κατάλληλη θεραπεία. Επίσης το έγγραφο αυτό ασχολείται με την μη παροχή συγκεκριμένης θεραπείας σε σε ε, μια συγκεκριμένη χώρα. Και εγώ εποφελούμαι από, τις, ε, από διασυνοριακή ε, περίθαλψη, γι' αυτό με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα αυτό. Και το άλλο θέμα είναι οι υπηρεσίε στι συνοριακέ περιοχέ, όπου είναι πολύ πιο εύκολο να, πάει, να μεταβεί κανεί σε άλλη χώρα για να ε, λάβει τη θεραπεία του ε, λόγω τη ε, ε πρόσβαση στι υπηρεσίε. Δεν θα πρέπει να ε, γίνουμε υπερβολικά γραφειοκρατικοί στο θέμα αυτό, διότι ο κόσμο που χρειάζεται ε, ιατρική περίθαλψη έχει ένα σωρό άλλα προβλήματα. Θα πρέπει λοιπόν να αποφύγουμε την υπερβολική γραφειοκρατία. Καταλαβαίνω ότι είναι απαραίτητη η προηγούμενη έγκριση, απ' την άλλη θα πρέπει να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία και θα πρέπει να επιδιώξουμε ε, να βρούμε να πετύχουμε την ισορροπία αυτή ε, φροντίζοντας οι, πληροφορίες, ε, οι απαραίτητες πληροφορίες να είναι διαθέσιμες στους παρόχους υπηρεσιών υγείας στα κράτη-μέλη και να μεταφέρονται στους ασθενείς. Επίσης, όταν κάποιος ε, μεταβαίνει σε άλλη χώρα για ε, ιατρική περίθαλψη, Θα πρέπει να φροντίσουμε ε, ε, το κράτος προέλευσης ε, να μην κλείνει την πόρτα, να μην λέει ότι «Α, συγγνώμη, πήγατε σε άλλη χώρα, πρέπει να και για την συνέχεια της θεραπείας να πάτε εκεί». Θα πρέπει δηλαδή να φροντίσουμε να υπάρχει σωστή ανταλλαγή πληροφοριών κάποιος Γερμανός πήγε στην ε, Ιρλανδία για ιατρική περίθαλψη. Οι γερμανικές αρχές όμως ε, δεν ήθελαν ε, να δώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες, να δώσουν το ιστορικό, διότι ο ασθενής πήγε σε ψυχιατρίο και θεωρείται ιατρικό απόρριτα. Ε, θα πρέπει δηλαδή να φροντίσουμε να διασφαλίσεται και η εμπιστευτικότητα, ε, να γίνεται όμως και σωστή ανταλλαγή πληροφοριών. Ε, ήταν μια συγκεκριμένη υπόθεση που προέκυψε, αλλά είναι ένα θέμα που έχει προκύψει αυτό της ανταλλαγής πληροφοριών. Είναι σημαντικό λοιπόν οι υπηρεσίε υγεία να ε, ε, συνεργάζονται μεταξύ του και επίση ω προ την συνέχεια τη θεραπεία, δηλαδή κάποιο που ε, λαμβάνει την κύρια θεραπεία σε άλλη χώρα αλλά πρέπει να παρακολουθηθεί η συνέχεια στο κράτο μέλο προέλευσή του, θα πρέπει να γνωρίζει ότι υπάρχει καλή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών των δύο χωρών. Επίση είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει νομική βεβαιότητα. Αυτό χρειάζεται να κάνουμε ε, στην οδηγία αυτή. Δεν ε, θα μπορέσουμε να απαντήσουμε σε όλα τα ερωτήματα. Ξέρω ότι η Επίτροπος εργάζεται σκληρά για να αντιμετωπίσει όλα τα ζητήματα. Ε, σε δύο-τρία χρόνια μπορεί να χρειαστεί να επανέλθουμε. Αλλά σημαντικό είναι να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Επικροτώ την πρόταση της ε, Επιτρόπου. Όλοι νομίζω μπορούμε να συμβάλλουμε στη βελτίωση του εγγράφου. Είναι σημαντικό όμως να πετύχουμε τη σωστή ισορροπία, διότι στο κάτω-κάτω τον ασθενή θέλουμε να φροντίσουμε. Και είναι σημαντικό να μην ε, κάνουμε υπερβολικά γραφειοκρατική τη διαδικασία, ώστε να εμποδίσουμε τους ανθρώπους ε, να λάβουν τη ιατρική περίθαλψη που χρειάζονται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ρούιλε. Η κυρία Γιώργενσεν. Δεν ξέρω, ε, ε, με την ηλικία θα το πάρουμε ή πιο όμορφη θα μιλήσει πρώτα. Ε, ή πιο άρρωστη. Θα μιλήσω δανέζικα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. ε, περίμενα εναγωνίως να εργαστώ πάνω στο θέμα αυτό, διότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους πολίτες της Ευρώπης και είμαι ευγνώμων προς την Επίτροπο που με την ανάληψη των καθηκόντων της αμέσως ξεκίνησε ε, να εργάζεται πάνω στο θέμα αυτό και έκανε πολύ καλή και ε, σωστή δουλειά για το θέμα αυτό η οδηγία αυτή και γενικά το θέμα ε, των διασυνοριακών ε, ε, υπηρεσιών υγείας είναι πολύ σημαντικό. Εγώ έχω μεγαλώσει στην Ήπεθρο. Εκεί συναντώ συχνά έναν ηλικιωμένο κύριο που οδηγάει το παπάκι του, έχει πίσω ένα ε, ε, μια κούτα στη σχάρα και πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζει. Ε, όλοι μας γνωρίζουμε τέτοιες φιγούρες και αυτόν σκέφτομαι με το συγκεκριμένο νομοθέτημα. Θέλω αυτός να έχει τη δυνατότητα να πάει στο εξωτερικό για να λάβει την απαραίτητη γιατρική περίθαλψη αν αυτό είναι απαραίτητο δεν έχει τις ίδιες δυνατότητες που έχουμε εμείς ε, που καθόμαστε εδώ σήμερα. Εμείς έχουμε χρήματα, ε, έχουμε τις δυνατότητες ε, και, και τις δυνάμεις να το κάνουμε αυτό και από ανθρώπινης και από οικονομικής πλευράς. Μπορεί να μην θέλει να το κάνει, αλλά πρέπει να έχει τη δυνατότητα να το κάνει και να μπορεί να διαλέξει εάν θέλει να πάει στο εξωτερικό μπορεί να έχει ένα εγγόνι πολύγλωσσο που να μπορεί να τον βοηθήσει. Ε, δεν θα πρέπει όμως ε, να, το αποκλείσουμε τις δυνατότητες. Θα πρέπει ο ίδιος να αποφασίσει αν θέλει να πάει στο εξωτερικό ή όχι. Ε, όπως καταλαβαίνετε από την εισαγωγή μου, με ενδιαφέρει να επικεντρωθώ στον ε, ασθενή και όχι στο σύστημα. Όταν όμως διαβάζω την πρόταση της ε, καλής συναδέλφου της κυρίας Βέρνο βλέπω ότι το σύστημα ε, βρίσκεται στο επίκεντρο. Εγώ δεν θέλω να διατηρήσω το σύστημα, θέλω να αλλάξω τα συστήματα προς όφελος του Ευρωπαίου πολίτη. Πρέπει να δημιουργήσουμε δυνατότητες ε, να φροντίσουμε να τηρούνται τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών ε, που θεσπίζονται με τη συνθήκη και που επιβεβαιώνονται από το ε, δικαστήριο. Από ό,τι καταλαβαίνω από την πρόταση της κυρίας Βερνιό, θέλει να οπισθοχωρήσει πολύ από την πρόταση της Κομισιόν και να ε, αντιταχθεί στις αποφάσεις του δικαστηρίου. Θέλει να υπερασπιστεί το σύστημα. Ως σκιώδης εισηγήτρια για την ομάδα των φιλελευθέρων επιθυμώ τα εξής Καταρχήν, η προηγούμενη έγκριση θα πρέπει να αποτελεί εξαίρεση, το επαναλαμβάνω, εξαίρεση. Διότι για τον άνθρωπο που σας μίλησα νωρίτερα που οδηγεί το παπάκι του στην εξοχή για να μπορεί να πάει στο εξωτερικό και να λάβει την απαραίτητη γιατρική περίθαλψη Πιστεύω ότι για τον άνθρωπο αυτό θα πρέπει η πληρωμή των υπηρεσιών να γίνει από το ένα σύστημα στο άλλο, από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Δεν θα πρέπει ο ίδιος να πρέπει να μπορεί να ε, προκαταβάλει το ποσό και να χρεωθεί για να λάβει μια ιατρική περίθαλψη σε κάποιο άλλο κράτος μέλος που είναι απαραίτητη για την επιβίωσή του. Εάν δεν φροντίσουμε τα χρήματα να βγαίνουν κατευθείαν από το ένα κράτο μέλο στο άλλο, τότε ε, οι άνθρωποι που δεν έχουν ε, πόρου ε, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν γιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό. Και θα πρέπει η υπηρεσία αυτή να είναι διαθέσιμη σε όλου του πολίτε τη Ευρώπη, όχι μόνο στου ισχυρού. Επίσης ε, θα πρέπει να υπάρχουν συστήματα πληροφόρησης, ε, συστήματα παροχής συμβουλών ε, τα οποία να λειτουργούν επαγγελματικά και σε πολλές χώρες διότι εάν θέλει κάποιος να έρθει στη Δανία δεν θα μπορεί ο καθένα να διαβάσει δανέζικα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό οι πληροφορίε αυτέ να παρέχονται σε περισσότερε γλώσσε. πέρα από την γλώσσα δηλαδή του, συγκεκριμένου κράτου μέλου. Τέταρτον, Θέλω ανεξάρτητα κέντρα πληροφόρησης που να μπορούν να συμβουλεύσουν τους ασθενείς στη ζούγκλα των ε, ιατρικών θεραπείων που προσφέρονται στα διάφορα κράτη-μέλη. Και ε, με την ε, ανεξάρτητη αυτή παροχή συμβουλών μπορεί να αποφασίσει ο ασθενής εάν θέλει να λάβει ε, γιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό. Είναι σημαντικό όμως η συμβουλευτική αυτή να είναι ανεξάρτητη, να μην αποτελεί μέρος του συστήματος, ενός συστήματος που έχει δικές του επιθυμίες σχετικά με τη γιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό. Ε, να μην ανήκει σε ένα σύστημα που ενδεχομένως λόγω οικονομικών προβλημάτων δεν θέλει να στείλει ασθενείς στο εξωτερικό. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό για μας τους φιλελευθέρους να υπάρχουν ανεξάρτητα κέντρα συμβουλών που να μπορούν να δίνουν σωστές ανεξάρτητες συμβουλές με αντικειμενική βάση ώστε ασθενής να μπορεί να λάβει απόφαση σχετικά με το αν επιθυμεί ή όχι να μεταβεί στο εξωτερικό για ιατρική θεραπεία. Η επιλογή όμως, η απόφαση θα πρέπει να είναι του ιδίου του ασθενή. Επίσης πιστεύω ότι είναι σημαντικό να έχουμε έναν Ευρωπαίο διαμεσολαβητή ασθενών ε, σε περίπτωση που υπάρχουν προβλήματα με την προηγούμενη έγκριση, με την ε, πληρωμή ε, της θεραπείας, θα πρέπει να μπορεί να παρέμβει τέσσερα πράγματα. Δηλαδή, η προηγούμενη έγκριση θα πρέπει ε, να είναι η εξαίρεση, η πληρωμή θα πρέπει να γίνεται κατευθείαν από το ένα σύστημα στο άλλο, από το, ε, από, το ε, ένα σύστημα στο άλλο. Ανεξάρτητα κέντρα πληροφόρησης και συμβουλευτικής και και ελπίζω η κυρία Βερνιό να ε, ε, ε, δεχτεί να μεταφέρει το επικεντρό της στον ασθενή. Τα συστήματα θα επιβιώσουν, θα επιβιώσουν αλλά πρέπει οι ασθενείς να επιβιώσουν και να έχουν εγκαίρως την σωστή γιατρική περίθαλψη. Δεν θα ήθελα να δω να συμβαίνει το αντίθετο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ρούιλε, ε, ναι, θα πρέπει να σκεφτούμε τον ασθενή και όχι το σύστημα και άκουσα το δικό σας ε, παράδειγμα με τον ε, ηλικιωμένο κύριο στην Ήπεθρο. Αυτός συνήθως θα μιλάει μόνο δανέζικα ή στη Γερμανία μόνο γερμανικά. Θα είναι πρόβλημα να ε, αποκτήσει εμπιστοσύνη σε έναν γιατρό που δεν μιλάει τη γλώσσα του. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτεί προσεκτικά εάν ε, θέλει να πάει στο εξωτερικό για ιατρική περίθαλψη, ε, διότι το κατόφλι αδοχή του είναι πολύ ψηλότερο από ό,τι άλλων. Αλλά υπάρχει το πρόβλημα για τον άνθρωπο αυτόν ότι στη Δανία γίνονται συνεχώς επενδύσεις στο γίνονται συνέχεια επενδύσεις στο ε, ε, σύστημα υγείας. Ε, ο άνθρωπος αυτός θα πρέπει λοιπόν να έχει την βεβαιότητα, την εμπιστοσύνη ότι το δανέζικο σύστημα θα συνεχίσει να επενδύει στο σύστημα υγείας και δεν θα βασίζεται στο, στην μετάβαση στο εξωτερικό των ασθενών. Ε, ρατώ γιατί η Επίτροπος έχει επιλέξει ως νομική βάση ε, το άρθρο 59 και όχι το άρθρο 152 παράγραφος 5 όπου αναφέρεται ε, σαφώς η ευθύνη των κρατών μελών και όπου αναφέρεται επίσης βιτά και η αρχή της επικουρικότητας. Θα ήθελα λοιπόν ως νομική βάση να έχουμε και το 152 όχι μόνο το άρθρο 59. Το πρώτο πρόβλημα. Δεύτερον, συμφωνώ με την προσέγγιση της κυρίας Βερνιό, αλλά θα ήθελα να αναφέρω ε, ένα ακόμα πρόβλημα. Ε, ας ξαναπάρουμε τον ε, γέρο αυτόν. Και αν αυτός προέρχεται από την Βουλγαρία ή από τη Ρουμανία, πόσοι ηλικιωμένοι άνθρωποι από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία θα μπορούσαν να έρθουν στην Γερμανία για ιατρική περίθαλψη χωρίς η Γερμανία να πει μέχρι η Γερμανία να πει ότι δεν αντέχει το σύστημά μας ε, ε, ε, να να περιθάλπει τόσους ασθενείς επειδή δεν είναι τόσο προηγμένα τα συστήματα υγείας στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία. Δεν μπορούμε λοιπόν να ανοίξουμε τα, τα συστήματα υγείας μας χωρίς να υπάρχει κάποια εξομοίωση των συστημάτων κάποια στιγμή θα συναντήσουμε το πρόβλημα αυτό και τίθεται το ερώτημα ποιος ε, μπορεί να εγγυηθεί ότι ε, θα ε, αναπτυχθούν τα συστήματα υγείας εάν δεν υπάρχει κάποιο ταμείο αντιστάθμισης, κάποιο ταμείο για την εξομοίωση, ποιοτική εξομοίωση των συστημάτων υγείας. Ε, χαίρομαι που η κυρία Βερνιό άρχισε να εξετάζει την πρόταση. Θα συνεχίσουμε την εξέταση, αλλά κατά τη γνώμη μου δεν είναι ακόμα έτοιμη η έκθεση αυτή για να την υιοθετήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Προτού να δώσω το λόγο στην Επίτροπο, θα ήθελα να επαναλάβω ε, τα συμπεράσματα του συμπεράσματος που ακούσαμε το 2004 ε, για τις ε, υπηρεσίες υγείας. From the Czech Could uh, Μήπως θα μπορούσατε να... Θα ήθελα... Θα ήθελα να μιλήσω τσέχικα, αλλά... Υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Όχι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τη διερμηνία. Μπορώ να μιλήσω τσέχικα. Ναι, βεβαίως. Ωραία. Θα μιλήσω τσέχικα. Ήθελα, όπως έλεγα, να σας ε, παρουσιάσω λίγο τα συμπεράσματα του σημεριναρίου που οργανώθηκε στις Βρυξέλλες για το θέμα αυτό. Είναι συμπεράσματα τα οποία υποστηρίζουν ε, ειδικοί ένα την Ευρώπη. Θα πρέπει να καθορίσουμε πάρα πολύ καλά το θέμα αυτό και μάλιστα με τρόπο που θα το κατανοούν και οι ασθενείς αλλά και όσοι είναι επαγγελματίε στον τομέα της υγείας για να μπορέσουμε να καθορίσουμε κατά πόσο κάποιος μπορεί να λάβει πρώτερη έγκριση για να ξέρει τι περίθαλψη μπορεί να του παρέχεται σε ένα κράτος μέλος. Είτε πρόκειται για νοσοκομιακή είτε πρόκειται για εξονοσοκομιακή περίθαλψη. Αυτά είναι συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν εμπειρογνώμονες στον τομέα αυτό. Επίσης θα πρέπει να δούμε και τι απαιτήσει υπάρχουν όταν θέλουμε να θεσπίσουμε ένα σύστημα ελέγχων και ασφάλειας στις υπηρεσίες υγείας. Θα πρέπει οι ασθενείς να έχουν μία σειρά αποδείκτες ασφάλειας για τις ε, υπηρεσίες περίθαλψης. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και για ποια χώρα μιλάμε σε κάθε περίπτωση. Επίσης, το κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να διασφαλίζει ότι θα έχει επαρκείς πληροφορίες για τους ασθενείς ως προς τις ε, δομές, ε, το χώρο ε, στον οποίο θα λάβουν περίθαλψη σε μια κάποια άλλη χώρα για να υπάρχει μια πανοραμική εικόνα των υπηρεσιών περίθαλψης που λαμβάνει αλλά και σε ποιες εγκαταστάσεις θα λάβει τέτοιες υπηρεσίες. Θα πρέπει να υπάρχει ισότητα και να είναι και ομογενείς οι υπηρεσίες περίθαλψης ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ο κανονισμός και υπάρχει και η νομολογία, μια σειρά αποφάσεις του δικαστηρίου, τις οποίες θα πρέπει να λάβουμε υπόψη, αλλά και να τις εναρμονίσουμε. Διότι όλα αυτά είναι υπέρ του πολίτη, υπέρ του ασθενούς. Ε, λέτε ότι έχουν δικαίωμα να λάβουν αποζημίωση για την παρήθελψη που τους ε, παρασχέθηκε και να λάβουν το ίδιο ποσό που θα λάμβαναν ε, στη χώρα τους. Διαπιστώσαμε για παράδειγμα ότι κάποιοι κατέβαλαν ε, ασφάλεια υγείας σε άλλη χώρα ε, και όχι στη χώρα διαμονής τους. Αυτά είναι παράλογα πράγματα και δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να γίνονται τα πράγματα ανεξέλεγκτα. Η κυρία Βερνιόν έλεγε ότι στο θέμα αυτό θα πρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ των επαγγελματιών ε, της υγείας και την κινητικότητα τη δική τους και την κινητικότητα των ασθενών. Κατά την άποψή μου, όντως, είναι 1% ο αριθμός των ασθενών που ε, εκμεταλλεύεται αυτή τη δυνατότητα μετακίνηση σε άλλη χώρα, αλλά πρόκειται για ένα ποσοστό το οποίο θα μέλλον θα αυξηθεί. Και επειδή ακριβώς θέλουμε να αυξήσουμε και την ποιότητα των υπηρεσιών ε, περίθαλψης, ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη και το θέμα από την απτική γωνία των ασθενών. Εγώ έκανα μία απόπειρα τον τελευταίο καιρό μέσω μια σειρά τροπολογιών ε, και σε άλλε επιτροπέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίω Επιτροπή ε, Γυναικών, να κάνουμε μια σειρά από για να εναρμονιστούμε λίγο και με τις αποφάσεις του δικαστηρίου. Να μην βρεθούμε ενώπιον μας κατάστασης ε, όπου θα εργαζόμαστε δεχόμενοι και πιέσεις και να καταλήγουμε σε πράγματα τα οποία δεν θα συνάδουν καθόλου με αυτά που αποφασίζει το δικαστήριο. Αυτά που είδαμε στις συζητήσεις του Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της Γαλλικής ε, Προεδρίας μας δείχνουν ότι οι ασθενείς ε, τελικά δείχνουν μια προτίμηση ε, σχετικά με την εξοικονόμηση δαπανών βραχυπρόθεσμα. Δηλαδή φαίνεται ότι οι ασθενείς αυτή τη στιγμή δεν έχουν πάρα πολύ καλές γνώσεις του θέματος και γνωρίζουν την κατάσταση από έξω προς τα μέσα. Δεν ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει πρέπει να μπορούμε να εφαρμόσουμε όλα όσα ακούσαμε σήμερα από τους συναδέλφους. Πολλές φορές οι πολιτικοί δεν μπορούν να δράσουν κατά των κυβερνήσεων των κρατών τους. Και τελικά δεν τους ενδιαφέρουν και καθόλου τα συμφέροντα των ασθενών. Στην πρώτη φάση είχαμε μία σειρά από σχόλια παρατηρήσεις. Τώρα θα ήθελα να ακούσουμε και πώς βλέπει η Επίτροπος τη σχέση μεταξύ της διαχείρισης ε, των υπηρεσιών υγείας και της κινητικότητας των ασθενών. Τι μπορούμε να κάνουμε σε επίπεδο συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών και επίσης θα ήθελα να ακούσω και τι έχετε να πείτε εσείς, διότι εμείς ως Επιτροπή εκτιμούμε ιδιαίτερα τα όσα κάνατε και εμείς εδώ βλέπουμε και πόσο καλύτερα δρούν οι γυναίκες σε σχέση με τους άντρες. Επιτρέψτε μου αυτό το σχόλιο, το οποίο είναι πολιτικά ίσως ε, ανορθόδοξο. Η Επίτροπος, παρακαλώ. Νομίζω ότι το τελευταίο σχόλιο δεν θα αρέσει ιδιαίτερα στους άνδρες συναδέλφους. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στα περισσότερα από τα σχόλιά σας. Ξεκινώντας από τον βασικό κανόνα ότι ο κανονισμός 1408 θα μείνει ανέγγιχτος και θα ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις για τις οποίες ισχύει τώρα. Επί παραδείγματι, Κάποιος από τους συναδέλφους σας αναφέρθηκε σε κατεπίγουσα περίθελψη. Εάν όντω κάποιο χρειάζεται κατεπηγόντω περίθελψη, τότε αυτό εμπίπτει στον κανονισμό 1408 και το κράτο μέλο είναι υπεύθυνο για την κάλυψη των δαπανών πλήρω. δεν θέλουμε να δώσουμε διέξοδο στα κράτη-μέλη για να αποφύγουν την εφαρμογή του 1408. Αυτό θα πρέπει σαφώς να αποτελεί προτεραιότητα. Μην ξεχνάμε όμως ότι υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις για τις οποίες το δικαστήριο είπε ότι πέραν των περιπτώσεων που εμπίπτουν στον κανονισμό, ο ασθενής έχει εγγενές δικαίωμα βάσει της συνθήκης να επιλέξει που θέλει να λάβει περίθελψη για τον οποιονδήποτε λόγο. Αυτό αποτελεί προσωπική απόφαση του ασθενούς και γι' αυτό ακριβώς και το δικαστήριο είπε ότι προκειμένου να ελέγχουμε το κόστος για το κράτος μέλος, τις περιπτώσεις τις οποίες ένας ασθενής αποφασίζει από μόνος του να μεταβεί στο εξωτερικό, τότε το κράτος μέλος θα πρέπει να πληρώνει μέχρι το κόστος που θα του αποζημιωνόταν στη χώρα του. Αυτή είναι η διαφορά. Τώρα, όσον αφορά σε αυτή την αναμενόμενη αύξηση της κινητικότητας των ασθενών μετά από την έγκριση της οδηγίας. Όντως υπάρχει περίπτωση να υπάρχει μια αύξηση. Σε αυτή την περίπτωση όμως, το δεκαστήριο πολύ σοφά είπε ότι πρέπει να προστατεύσουμε τα εθνικά συστήματα υγείας, δίνοντάς τους το δικαίωμα να εφαρμόσουν τον κανόνα της πρώτερης έγκρισης. Η πρώτερη έγκριση όμως δεν είναι κάτι που επινοήσαμε εμείς. Το δικαστήριο είπε κάντε μία διάκριση μεταξύ πρώτερης έγκρισης για μη νοσοκομιακή περίθαλψη, για την οποία δεν θα πρέπει να ισχύει, και αυτό το λέει πάρα πολύ σαφώς, και της πρώτερης έγκρισης για νοσοκομιακή περίθαλψη, εάν αυτή είναι απαραίτητη και εφαρμόζεται αναλογικά. Αν ένας ασθενής λοιπόν έχει έρθει από την αρχή και πει ότι Φοβάμαι, συγγνώμη, αν ένα κράτο μέλο έρθει από την αρχή και πει ότι φοβάμαι ότι θα έχω αύξηση και θα εφαρμόσω από την αρχή τον κανόνα τη πρώτερη έγκριση, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά το ίδιο το δικαστήριο είναι που θα το κηρύξει αυτό παράνομο. Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το δικαστήριο θα σα πει ότι είναι παράνομο. Το δικαστήριο σαφώς λοιπόν είπε ότι αν θεωρείται απαραίτητο για την προστασία των εθνικών συστημάτων και είναι αναλογικό και εφαρμόζεται χωρίς καμία διάκριση. Οι δύο τομείς ε, στους οποίους νομίζω ότι θα έχουμε αύξηση είναι στα σύνορα, στις περιπτώσεις που θα έχουμε στα σύνορα, το οποίο θα είναι πολύ πιο πρακτικό για κάποιον ασθενή να πάει στην ε, διπλανή χώρα και να λάβει περίθαλψη και στην περίπτωση των σπάνιων ασθενών, εκεί όντως λογικά προβλέπω ότι εάν ένας ασθενής πάσχει από μια σπάνια νόσο για την οποία δεν υπάρχει περίθαλψη στη χώρα του, θα αποφασίσει να μεταβεί σε κάποιο ιατρικό κέντρο στο εξωτερικό για να λάβει θεραπεία. Και αυτό άλλωστε θα είναι και το προστιθέμενο όφελος για τον ασθενή και γι' αυτό ακριβώς έχουμε και αυτή την διάταξη για συνεργασία μεταξύ κέντρων αναφοράς διότι υπάρχουν, ε, υπάρχει πληθώρα σπάνιων ασθενειών και θα είναι αδύνατο τα κράτη-μέλη να οργανώσουν τα εθνικά συστήματα υγεία τους με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να καλύψουν όλες αυτές τις ε, σπάνιες νόσους που αριθμούν περίπου μεταξύ 5 και 7 χιλιάδων. Τώρα, πληροφόρηση και η ποιότητα της είναι νομίζω τα δύο πρόσθετα στοιχεία τα οποία προσδίδουν αξία σε αυτή την οδηγία διότι όπως πολύ σωστά επισημάνατε κι εσείς θα πρέπει να προσέξουμε τον ασθενή και όχι το σύστημα. Πρέπει να δούμε πώς το σύστημα μπορεί να εξυπηρετήσει τον ασθενή. Είναι λοιπόν ικανή και αναγκαία συνθήκη να δώσουμε στον ασθενή όσο το δυνατόν περισσότερε πληροφορίε και αυτέ οι πληροφορίε θα πρέπει να είναι συμπεφωνημένε μεταξύ των κρατών μελών ώστε κατά την τελική του ανάλυση να υπάρχει ένα δίκτυο σημείων επαφή το οποίο θα επιτρέπει να αποφασίσουν, να συμφωνήσουν μεταξύ τους ποιες πληροφορίες θα πρέπει να ανταλλάσσουν. Επίσης, αυτό που ζητάμε από τα κρατη να, από τα κράτη να κάνουν ως προς την ποιότητα και την ασφάλεια είναι να θεσπίσουν πρότυπα για την ποιότητα και την ασφάλεια, προδιαγραφές. Δεν τους ζητάμε να εναρμονίσουν τα συστήματά τους, ούτε να έχουν ε, ε, ε, κράτη-μέλη που ήδη έχουν προδιαγραφές να εφαρμόσουν άλλες προδιαγραφές. Αρκεί να μας πούνε ότι εφαρμόζουμε χι προδιαγραφές και εποπτεύουμε την εφαρμογή αυτών των προδιαγραφών. Αυτό μόνο ζητάμε από τα κράτη-μέλη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον ασθενή πριν φύγει από τη χώρα του να ξέρει τι τον περιμένει, τι θα λάβει και να είναι καθησυχασμένος ότι θα έχει την ποιότητα και την ασφάλεια που χρειάζεται για την υγεία του. Και αυτό είναι κάτι το οποίο χρειάζεται ένας ασθενής προκειμένου να λάβει μια ενημερωμένη απόφαση. Όσον αφορά τώρα την προκαταβολή των δαπανών. Κανένας δεν μιλάει για προκαταβολή. Δεν υπάρχει τίποτα λοιπόν στην οδηγία που να απαγορεύει σε ένα κράτος μέλος να ε, συζητήσει με κάποιον ο οποίος παρέχει περίθαλψη στο εξωτερικό για να κάνει μια άμεση πληρωμή. Αυτό σαφώς θα εξυπηρετήσει τον ασθενή και είμαστε υπέρ του, αλλά εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα να το ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη είναι ελεύθερα να το κάνουν αν θέλουν. Ε, regarding για την νομική βάση. Αυτό δεν ήταν πολιτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι φυσική απόρρια των αποφάσεων του δικαστηρίου, διότι οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αφορούν τις ελευθερίες της ενιαίας αγοράς βάσει του άρθρου αυτού. Το άρθρο 152 ναι μεν έχει μεγάλη σχέση με το θέμα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα μας δώσει τη δυνατότητα να βασίσουμε μια οδηγία τέτοια υφής ε, στο άρθρο αυτό, το 152. Το αναφέρουμε φυσικά στην οδηγία και θα το σεβαστούμε το άρθρο αυτό, διότι λέμε πολύ συγκεκριμένα στην οδηγία ότι σεβόμαστε το δικαίωμα των κρατών μελών να οργανώσουν τα συστήματα υγείας τους όπως φρονούν ότι πρέπει να τα οργανώσουν για να δώσουν στους ασθενείς ε, τα ωφέλη που θέλουν να τους δώσουν και να προσφέρουν στους ασθενείς ε, τα φάρμακα που θα αποφασίσουν. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε τίποτα περισσότερο από τα κράτη-μέλη. Η ανταλλαγή πληροφοριών είναι πάρα πολύ σημαντική συμφωνώ και εγώ και υπάρχει και συγκεκριμένη διάταξη στην οδηγία για το θέμα αυτό, διότι όταν ένας ασθενής πηγαίνει στο εξωτερικό και μετά επιστρέφει στη χώρα του για την ε, παρακολούθηση, είναι απαραίτητο να διασφαλίσουμε το δικαίωμα αλλά και το καθέγον των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας να ανταλλάσσουν πληροφορίες. Όλες τις πληροφορίες που έχουν για τον ασθενή τους σεβόμενοι φυσικά και τα όσα αφορούν το προσωπικά δεδομένα και το σεβασμό τους. rightly. Κάποιοι από εσά πολύ σωστά αναφερθήκατε σε δύο πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Τις υφιστάμενες ανισότητες και ε, ε, able and number of health το πόσο σημαντικό είναι να έχουμε ικανούς ε, επαγγελματίες στον τομέα της υγείας αλλά και επαρκή αριθμό επαγγελματιών. Διότι η βάση της πυραμίδας είναι όντως η, τα ιατρικά επαγγέλματα. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως σα είπα, δημοσιεύσαμε τον περασμένο Δεκέμβριο μια πράσινη βίβλο για το εργατικό δυναμικό στον τομέα της υγείας και έχουμε ξεκινήσει μια διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερομένους για να διαπιστώσουμε πώς μπορούμε να καλύψουμε αυτές τις απαιτήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, κυρίως βάσει των ανισοτήτων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή μεταξύ δυτικών και ανατολικών κρατών και την κινητικότητα των επαγγελματιών αυτών και επίσης κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και κάποια κράτη-μέλη ήδη το χρησιμοποιούν έχουμε δώσει περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ στα διαρθρωτικά ταμεία 5 εκατομμύρια δις, συγγνώμη, στα διαρθρωτικά ταμεία για να μπορέσουμε σταδιακά να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να φτάσουν σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο παροχής ε, περίθαλψης. Αυτό είναι στο πρόγραμμα εργασίας ε, το δικό μου και του Επιτρέπου Σπίτλα και θέλουμε να έχουμε μια ανακοίνωση αργότερα εντός του έτους για να δούμε πώς μπορούμε να καλύψουμε αυτές τις ανισότητες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι ναι, συμφωνούμε και εμείς, είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό και ως προϋπόθεση για να πείσουμε τους ασθενείς να μείνουν στη χώρα τους και να μην ε, γυρνάνε σε όλη την Ευρώπη. Έχω σημειώσει όλα σας τα σχόλια, πέραν αυτών που σχολίασα και θα τα λάβω φυσικά υπόψη όταν θα κάνουμε την αναθεώρηση και θα έχουμε την τελική εκδοχή της οδηγίας μας. Σας ευχαριστούμε. Έχουμε ακτου, ακόμα οκτώ μιλητές. Η κυρία Σέντερσολτ έχει πρώτο λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε Βασιλείου και σε εσά εύχομαι καλή χρονιά και εγώ με τη σειρά μου. Καταλαβαίνουμε ότι έχετε αρκετά δύσκολα θέματα να αντιμετωπίσετε στο άμεσο μέλλον και ελπίζω το Κοινοβούλιο στο μέλλον σας διευκολύνει περισσότερο από ό,τι έχει κάνει ως τώρα. Οι πρόσφατες εξελίξεις στα θεσμικά όργανα φαίνεται να έχουν διακυβεύσει κάποιες από τις ενέργειες των κρατών μελών που ε, οργανώθηκαν από την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. ο σχεδιασμός της πρώτερης έγκρισης καθόλου δεν βλέπω να ευθυγραμμίζεται με την ε, νομολογία. Θα σήμαινε ότι μια με επίσκεψη ρουτίνα στον οφθαλμίατρο θα απαιτούσε πρώτερη έγκριση. Εάν δείτε τις τροπολογίες για τα άρθρα 7 και 8 και πώς έχει η κατάσταση για τους ασθενείς στην πραγματικότητα, θα αντιληφθείτε ότι δεν οδηγούμαστε έτσι σε νομική βεβαιότητα. Η Επιτροπή ΙΜΚΟ και το Κοινοβούλιο ζήτησαν κωδικοποίηση της ε, υπάρχουσας νομολογίας. Ελπίζω ότι θα γίνει κάποια στιγμή αυτό, αλλά σίγουρα αυτή, ακόμη δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο με την πρόταση αυτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι θεματοφύλακα των συνθηκών και προασπίζεται τα συμφέροντα των πολιτών. Γι' αυτό και έχω ένα συγκεκριμένο ερώτημα για σας. Θα αποσύρει η Επιτροπή ολόκληρη την πρόταση για την κινητικότητα των ασθενών ή μέρο τη, εάν τα δικαιώματα των ασθενών βάσει του υπάρχοντος κεκτημένου δεν καλύπτονται τελικώς. Uh, Σημαντικό σχόλιο. Κυρία Κέμπχαρτ έχει ζητήσει το λόγο. Ähm, Ευχαριστώ. Έχει περάσει η ώρα, γι' αυτό θα είμαι σύντομη. Έχουμε και τις ψηφοφορίες που μας περιμένουν. Καταρχάς, η περίθαλψη, οι υπηρεσίε οικονομική περίθαλψη είχαν ε, ξερεθεί από την ε, οδηγία για τι υπηρεσίε. Είχαμε πει ότι το τομέα τη υγεία είναι ένα τομέα με πολλέ ιδιαιτερότητε που δεν μπορεί να καλύπτεται από τα εμπορικά ζητήματα. Γι' αυτό. Γι' αυτό γιατί περιλαμβάνει ασθενεί, περιλαμβάνει καταστάσει που μπορεί να ενέχουν και εξάρτηση από τον παρέχοντα μια υπηρεσία. Θυμάμαι αυτό το παράδειγμα της κυρίας ε, Γιόγκινσεν, αυτό που μας έλεγε προηγουμένως, τον κύριο αυτό που πάνω στο παπάκι του αναγκάζεται να οδηγεί στην εξοχή και έχει δίκιο. Έχει δίκιο γιατί θα πρέπει να μπορεί να λάβει ιατρική περίθαλψη κοντά στον τόπο κατοικίας του. Θα πρέπει να μπορούν οι Ευρωπαίοι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας. Και έχετε δίκιο και εσείς βεβαίως ότι υπάρχουν ασθενείς που θα πάνε στο εξωτερικό εάν ε, πιστεύουν ότι χρειάζεται να λάβουν περίθαλψη αλλού ή κατά τη διάρκεια των διακοπών τους λόγου χάρη. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να επιληθούν. Γι' αυτό η οδηγία αυτή ούτως ή άλλως είναι σημαντική. Αλλά κατά τα άλλα να πω ότι μου φάνηκε κάπως περίεργο το γεγονός ότι η οδηγία αυτή τελικά πάει κάπως μακριά. Δηλαδή, πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει με την νομική βάση. Εδώ δεν συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, κυρία Επίτροπε. Κατά την προηγούμενη θητεία συμμετείχα στην ε, Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και ήμουν εισηγήτρια για το θέμα αυτό της νομικής βάσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν το συζητήσαμε αυτό το θέμα της νομικής βάσης μας έλεγε ανέκαθεν για την ειδική περίθαλψη Θα έπρεπε να τρέξουμε στο άρθρο που αρμόζει. Και είχαμε κοιτάξει το άρθρο 95 για την εσωτερική αγορά και το 158 που αφορά τα θέματα υγείας και προσπαθήσαμε να είμαστε συνεπείς σε σχέση με όσα γίνονται ω τώρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως γιατί δεν χρησιμοποιούμε κάτι τέτοιο και τώρα στο 152 υπάρχει και η επικουρικότητα και ο σεβασμός των εθνικών συστημάτων, αλλά υπάρχει και παραπομπή στο άρθρο 95. Νομίζω ότι θα ήταν ιδανική επιλογή το 152 για νομική βάση. Θα ήταν πολύ καλή επιλογή και θα ήταν και ξεκάθαρα τα πράγματα για τον Ευρωπαίο πολίτη. Θα πρέπει Επίση, να δούμε τι γίνεται με τι αποφάσει του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που έχει αρμοδιότητα να αποφανθεί για θέματα υγεία και διαφορέ τέτοιου είδου. Το Κοινοβούλιο αποφάσισε σε κάθε περίπτωση ότι εδώ προτεραιότητά μα δεν πρέπει να είναι η εσωτερική αγορά, αλλά τα δικαιώματα των ασθενών. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή τη συζήτηση πρέπει σαφώ να την ολοκληρώσουμε. Ναι. Σαφώς η κοινωνική διάσταση μας ενδιαφέρει και η περίπτωση των εργαζομένων σαφώς. Ο κύριος Μπούς. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρία Επιτροπέ, θέλω να σας συγχαρώ για την εξαιρετική και πολύ πιστική σας παρέμβαση. Είναι πολύ σημαντικό να συζητήσουμε την κινητικότητα των ασθενών και να θυμόμαστε ότι σήμερα 1% των Ευρωπαίων πολιτών αναζητούν περίθαλψη στο εξωτερικό. Και είναι πολύ περισσότεροι πολίτες που στο μέλλον θα, θα αναζητήσουν τέτοιες υπηρεσίες στο εξωτερικό. Εκτός και αν δώσουμε πολύ καλά κινήτρα στα εθνικά συστήματα υγείας για να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους και το πόσο προσβάσιμα είναι. Πάντως, νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση οι ασθενείς θα προτιμούν να λαμβάνουν ε, στη χώρα τους περίθαλψη παρά στο εξωτερικό, αρκεί όμως τα συστήματα να είναι καλής ποιότητας. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει σαφώς αποφασίσει ήδη ότι τα δικαιώματα των πολιτών ε, πρέπει να προστατευτούν και αυτό που μας έχει αναθέσει είναι να δούμε εμείς τις λεπτομέρειες του πώς θα υλοποιήσουμε αυτή την προστασία των δικαιωμάτων ασθενών. Ελπίζω ότι οι ενώσει ασθενών ε, και όλοι οι θυνοντές θα ασκήσουν πίεση στις κυβερνήσεις για να αποδεχτούν αυτή την πρόταση και νομίζω η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει σοβαρά την ιδέα να οργανώσει κάποια ενημερωτική εκστρατεία στα κατημέλη προκειμένου να εξηγήσει στους πολίτες ποια είναι τα ωφέλη αυτής της πρωτοβουλίας. Ευχαριστώ. Thank you very much. And ε, Mrs. Ευχαριστούμε κυρία Σάλντεμόζα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή σας παρουσίαση. Ένα μικρό σχόλιο και θα θέλω να ξεκινήσω με αυτό. Συζητούμε σαν να υπάρχει διαφορά μεταξύ των δικαιωμάτων των αστερών από τη μια και τη διατήρηση καθώ και βελτίωση των εθνικών συστημάτων υγεία από την άλλη. Δεν θα έπρεπε να κάνουμε μια τέτοια εσφαλμένη διχοτόμηση μεταξύ των ε, ασθενών και των συστημάτων υγεία. Μα ενδιαφέρει ο πολιτικό σχεδιασμό εδώ. Τι μέθοδο θα χρησιμοποιήσουμε για να, για να βεβαιωθούμε ότι όλοι οι ασθενεί θα λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή περίθαλψη. Μην κάνουμε λοιπόν εσφαλμένε συγκρίσει. Τώρα, πέραν αυτού, να πω ότι Ανησυχώ λίγο για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η πρόταση στις ανισότητες μεταξύ παλαιών και νέων κρατών μελών. Ως πολίτης ε, παλαιού κράτους μέλους, πρέπει να πω ότι η περίθαλψη κοστίζει πολύ στη Δανία. Πολλές φορές λοιπόν φεύγουν στο εξωτερικό για περίθαλψη αλλού στην Ευρώπη. Οι πολίτες της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας όμως δεν μπορούν να κάνουν το ίδιο χωρίς να δουν το κόστος να πολλαπλασιάζεται Άρα ανησυχώ λίγο κατά τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η πρόταση αυτή, διότι δεν θέλουμε να έχουμε διακριτική μεταχείριση των πολιτών. Θα μπορούσατε να μα πείτε λίγα λόγια για το τι σκοπεύετε να κάνετε για να γεφυρώσετε αυτά τα μεγάλα χάσματα ενδεχομένω. Ευχαριστούμε η κυρία Πλεστίνσκα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κυρία Επιτροπέ για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας. Ήθελα στα σχόλια των προηγουμένων να προσθέσω το εξή. Είναι πολύ σημαντικό να οργανωθεί κάποια ενημερωτική εκστρατεία εδώ. Να πούμε ότι ένας λόγος που οι ασθενείς δεν ανατρέχουν στη διασυνοριακή περίθαλψη είναι επειδή δεν υπάρχει επαρκή πληροφόρηση, μπορεί να έχουν κακέ εμπειρίες σε περίπτωση που κατεπηγόντω χρειάστηκαν θεραπεία ή περίθαλψη αν είχαν κάποια τύχημα στο εξωτερικό και επίσης υπάρχει και άνεση χρηματοδότηση. Στην Σλοβακία λόγου χάρη ε, το κόστος της περίθαλψης ε, είναι πολύ ψηλό, ειδικά το τελευταίο διάστημα ειδικά με την προσχώρησή μας στην Ευρωζώνη. Οπότε θα πρέπει να σκεφτούμε αυτό πώς μπορεί να επηρεάσει τις διαφορές μεταξύ κρατών μελών και να φροντίσουμε να μην υπάρξει διακριτική μεταχείριση. Και είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι γίνεται και με συγκεκριμένε υπηρεσίε. Οδοντιατρικέ υπηρεσίε, λόγω χάρη, που σε μια συγκεκριμένη χώρα μπορεί να είναι καλή ποιότητα και κάποιοι να προτιμούν ούτω ή άλλω να πηγαίνουν στη χώρα αυτή. Επίση, υπάρχουν και γλωσσικοί φραγμοί. Μπορεί να χρειάζονται διορθώσεις ή επεμβάσεις ε, της ηλεκτρονικής οδού, ώστε να αποφεύγουν ε, οι ασθενείς το να ανατρέχουν ε, σε μεταφράσεις των εγγράφων και των χαρτιών που πρέπει να δώσουν στους γιατρούς. Ο κύριος Αγγελάκας για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος με τέσσερις συγκεκριμένες τοποθετήσεις, αναφέροντας και τα άρθρα. Έχω την αίσθηση, κυρία Επίτροπε, ότι ακόμα δεν είναι εξαιρετικά ε, σαφές στο άρθρο 8 τι εννοούμε νοσοκομιακή περίθαλψη και τι εξονοσοκομιακή. Τα διάφορα συστήματα υγείας στα διάφορα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικούς χαρακτηρισμούς. Αυτό θα προκαλέσει σύγχυση. Κάπως πρέπει να το δείτε. Για το θέμα δεύτερον της αναγνώρισης των φαρμακευτικών συνταγών σας έχω ξαναρωτήσει και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Κράτη-μέλη έχουν θετική λίστα, κράτη-μέλη έχουν αρνητική λίστα, κράτη-μέλη δεν έχουν λίστα φαρμάκων, θα δημιουργηθεί σύγχυση. Άρθρο 8 παράγραφος Β. Μιλάτε για έναν κατάλογο ασθενειών που θα είναι επιλέξιμες και λέτε ότι το κριτήριο είναι η πολύ εξειδικευμένη ή δαπανηρή ιατρική υποδομή. Και αυτό είναι κάπως ασαφές. Για ένα κράτος μέλος μια υποδομή ιατρική μπορεί να είναι ε, δαπανηρή, για ένα άλλο όχι. Εξαρτάται από το επίπεδο υγείας. Πρέπει να το δούμε. Και τελευταία παρατήρηση και κλείνω. Στο άρθρο 20 μιλάτε για μια έκθεση πρόδρου λειτουργίας της ε, οδηγίας μετά από πέντε χρόνια. Προσωπική μου γνώμη είναι ότι είναι πολύ μεγάλο διάστημα για να μπορέσουμε να δούμε τι δεν πήγε καλά και τι πήγε καλά για να το διορθώσουμε. Μήπως έπρεπε να γίνει αυτό μια διετία ή τριετία για να δούμε πώς πηγαίνουμε. Ευχαριστώ. ευχαριστώ κύριος Σουάπ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Έχουμε εδώ σημαντικό πολιτικό πρόβλημα. Η όλη συζήτηση δείχνει ότι δεν θέλουμε να ασχοληθούμε με τον πυρήνα του προβλήματος. Κυρία Επίτροπε, βρίσκεστε υπό σημαντική ε, πίεση από τα κράτη-μέλη που ε, κρύβονται πίσω από την αρχή της επικουρικότητας και, διάφορες παραγράφους, ε, και διάφορα άρθρα ε, των συνθήκων και θέλουν λοιπόν να διατηρήσουν όσο γίνεται περισσότερη ανεξαρτησία. άσχετα λοιπόν το πιο άρθρο της συνθήκης λοιπόν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως νομική βάση είναι πολιτικό θέμα. Τελικά όμως μάλλον θα πρέπει να καταλήξουμε στο ε, άρθρο 152 διότι κυρία Κέπχαρτ έχετε δίκιο ή είναι αυτή η σωστή νομική βάση. Αλλά αν ξεκινούσαμε από εκεί δεν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε καθόλου. Ε, κυρία Ρίλε και κυρία Ρίς Γιάνσον, όσον αφορά την ε, ισότητα των ε, φύλων, ε, μήπως θα έπρεπε τον ηλικιωμένο κύριο από τη Δανία τη Γερμανία να τον στείλουμε σε κάποια νεαρή κυρία στην ε, Ισπανία. Ε, μόνο το 1% των ε, πολιτών έχουν τη δυνατότητα ή τη θέληση να κάνουν χρήση διασυνοριακών υπηρεσιών υγείας. Οπότε, ναι, δεν βρίσκω τη συζήτηση τελείως αδικαιολόγητη, τη βρίσκω όμω πολύ υπερβολική. Στην ε, Ρώμη, για παράδειγμα, υπάρχει ειδικό κέντρο για ε, τους καρκίνους ε, του δέρματος. Αλλού υπάρχουν ειδικά κέντρα για, τις, για τον καρκίνο του προστάτη. Υπάρχουν κάποιες, κάποια τέτοια κέντρα βάρους, αν το θέλετε, αλλά πέρα από αυτό ε, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αλλάξουμε ε, τους εθνικούς κανόνες για την ευθύνη των ε, γιατρών για τους λόγους αυτούς. Ούτως ή άλλως είναι πολύ, ιδιαίτερα πολύπλοκα τα θέματα αυτά για τους ασθενείς. Νομικός είμαι και εντός της Γερμανίας υπάρχουν, εκκρεμούν υποθέσεις ευθύνη γιατρών, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποδείξει κανείς τελικά ποιος γιατρός έκανε λάθος. Ε, ε, νομίζω λοιπόν ότι δεν πρέπει να αλλάξουμε τους κανόνες για την ευθύνη των γιατρών. Ε, αυτό θα πρέπει να το αφήσουμε στην επικουρικότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την τελευταία, παρατήρηση, την τελευταία παρέμβαση την έχει ο κύριο Σμιτ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω την Επίτροπο. Νομίζω ότι η Επιτροπή πράγματι χρειαζόταν ε, μια θαραλέα γυναίκα ε, που, ε, για να υποβάλει την πρόταση αυτή. Έχω ένα ερώτημα σχετικά με το χρονοδιάγραμμα. Άκουσα τη συζήτηση. Ασχολούμαι με την, ε, τις υπηρεσίες υγείας σε περιφερειακό επίπεδο στην πατρίδα μου από το 1985 και με εκπλήσει που ακούω τους συναδέλφους να δημιουργούν νέα εμπόδια. Επιτέλους ε, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου ε, το Κοινοβούλιο μπορεί να ε, ξαναφτάσει κοντά στους πολίτες. Οι υπηρεσίες υγείας βρίσκονται κοντά στην καρδιά του κάθε πολίτη και σε πολλά από τα κράτη-μέλη μας υπάρχουν ουρές, ουρές. Ο κόσμος περιμένει μήνες και χρόνια για υπηρεσίες υγείας. Αν ήμουν πολιτικός στη Γαλλία όπου το 54% ε, των πολιτών θέλουν να, πάνε, να εγκαταλείψουν τη Γαλλία και να πάνε αλλού για υπηρεσίε ε, υγεία, θα έκανα κάτι γι' αυτό. Εγώ μένω 20 λεπτά από τη Δανία. Είναι πολύ δύσκολο να πάνε οι Σουηδοί ε, στη Δανία. Ναι, εντάξει, θέλουν να πάνε για τι μπύρε, αλλά για τι υπηρεσίε υγεία είναι πολύ δύσκολο να πάνε. Θέλουν να βρίσκονται στην πατρίδα του. Η πεθερά μου έπρεπε να πάει εκατοντάδες ε, χιλιόμετρα ε, για να πάει σε καλό χειρουργείο. Δεν ήθελε να το κάνει αυτό, ήθελε να χειρουργηθεί κοντά στο σπίτι της. Να μην υπερβάλλουμε τα προβλήματα. Εάν όμως είναι να κάνουμε κάτι θα πρέπει να το κάνουμε σε αυστηρό νομικό πλαίσιο. Νομίζω ότι η Επίτροπος βρίσκεται σε καλό δρόμο, θα είναι δύσκολο. Ε... Μπορεί να μην έχετε πολλή υποστήριξη από το Κοινοβούλιο μας, από τους πολίτες πάντως σίγουρα θα έχετε. Και η ερώτησή μου, τι γίνεται με το χρονοδιάγραμμα. Πότε πιστεύετε ότι μπορεί το θέμα αυτό να υποβληθεί στο Συμβούλιο. Φέτος το φθινόπωρο. Πότε πιστεύετε, διότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να ενεργήσετε γρήγορα. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία, κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ για την ε, πολύ ε, σωστή τελική σας παρατήρηση. Κύριε Επίτροπε, έχετε πέντε λεπτά μόλις ε, για να μας πείτε τα βασικά. Ε, ποιο είναι το μήνυμά σας. Ευχαριστώ. Μου τέθηκε ένα πολύ δύσκολο ερώτημα. Μόλις πριν κάνα δύο μήνες ξεκινήσαμε. Και τώρα με ρωτάτε αν είμαι διατεθειμένη να ανακαλέσω. Όχι. Είμαι αποφασισμένη να συνεχίσω διότι πιστεύω ότι το χρωστάμε στους ασθενείς. Άσχετα από το τι πούμε εδώ, άσχετα από το τι λέει το Συμβούλιο, υπάρχουν τα δικαιώματα των ασθενών που θεσπίζονται στη συνθήκη Και όσο περισσότερο το συζητάμε, τόσο περισσότεροι θα εγκαταλείψουν τη χώρα τους να πάνε σε άλλη χώρα για ε, περίθαλψη χωρίς ε, ασφάλεια, χωρίς βεβαιότητα και πιστέψτε με μόνο ε, όσοι έχουν τα χρήματα να πληρώσουν δικηγόρο για να πάνε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα μπορέσουν να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους και δεν το θέλουμε αυτό διότι αυτό πραγματικά δημιουργεί ανισότητα. Έχουμε λοιπόν χρέος να προχωρήσουμε. πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αυτά εξαρτάται από εσά, του ευρωβουλευτέ. Από εσά εξαρτάται. Εάν καταφέρουμε να ολοκληρωθεί η πρώτη ανάγνωση πριν το τέλος της θητείας σας, αυτό θα είναι πολύ χρήσιμο και πολύ θετικό. Όλα εξαρτώνται από εσά τους ευρωβουλευτές. Η κυρία Βερνιό ανέφερε το 54% των ε, ανθρώπων που θέλουν ιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό. Με όλο το σεβασμό, δεν νομίζω ότι λένε ότι θα ήθελαν να πάνε στο εξωτερικό. Θα ήταν διατεθειμένοι να πάνε αν ήταν απαραίτητο, νομίζω. Ε, είναι κάτι διαφορετικό αυτό. Εάν όμως ρωτήσετε τον οποιοδήποτε πολίτη στο δρόμο, ε, είσαστε διατεθειμένοι να πάτε εάν ε, έχετε τη δυνατότητα, φυσικά θα πούνε ναι. Ποιος δεν θέλει να ταξιδέψει. Εάν όμως τους δώσουμε τις πληροφορίες, τι έχουν να περιμένουν, τι θα λάβουν ως αποζημίωση, επιστροφή των εξόδων το, την κούραση του ταξιδιού, τις δυσκολίες της γλώσσας, ε, τις δυσκολίες του να είναι κανείς ε, μόνος του σε ξένη χώρα. Πιστέψτε με το 54% αυτό θα είναι πολύ μικρότερο ποσοστό τελικά. Είναι πολύ δύσκολο το θέμα των υπηρεσιών υγείας, ε, το εξετάζουμε προσεκτικά και ελπίζω ότι εσείς οι Ευρωβουλευτές ε, θα συμμετάσχετε στην ε, συζήτηση για την Πράσινη Βίβλο και θα μας βοηθήσετε έτσι. Προσβλέπουμε στην καλή συνεργασία μαζί σας. Ο κύριος Αγγελάκας ανέφερε τρία πολύ σημαντικά θέματα. Την αμοιβαία αναγνώριση των γιατρικών συνταγών. Έχουμε κανόνες ενισχύει που είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν. Με την οδηγία αυτή θέλουμε με την διαδικασία της επιτροπολογίας να ορίσουμε μια σειρά εμπειρογνωμόνων που θα εξετάσουν πώς μπορούμε να διευκολύνουμε τα φαρμακεία, τους γιατρούς κλπ. για να διευκολύνουμε τελικά τους ε, ασθενείς. Βρισκόμουν στην, ε, στο Λονδίνο την προηγούμενη εβδομάδα, μίλησα με τους ανθρώπους από την ΕΜΕΑ και τους ρώτησα είναι δυνατόν να έχουμε έναν κοινό κατάλογο φαρμάκων σε όλη την Ευρώπη. Αυτό θα μας διευκόλυνε πάρα πολύ. Έχουν πρόβλημα. Χρειάζονται στοιχεία από τα κράτη-μέλη δεδομένα που είναι πολύ δύσκολο ε, να δώσουν τα κράτη-μέλη, πολύ ακριβό να τα συλλέξουν και ε, εάν δεν έχουν τα στοιχεία αυτά, και έχουν ξεκινήσει και έχουν ξεκινήσει καλά, αλλά εάν δεν λάβουν τα ε, δεδομένα αυτά από τα κράτη-μέλη, δεν θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους. Στόχος μας είναι με την οδηγία αυτή να διευκολύνουμε τη συγκεκριμένη διαδικασία. Αναφερθήκατε στην πενταετία αναθεώρηση. Δεν επιμένουμε αυστηρά στη πενταετία. Υπολογίζουμε όμως ότι με την υιοθέτηση της οδηγίας, με τη διαδικασία της επιτροπολογίας θα πρέπει να ληφθούν κάποιες αποφάσεις και αυτό θα πάρει χρόνο. Μέχρι να τεθεί σε ισχύ η οδηγία αυτή θα περάσει χρόνος. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η πενταετία είναι λογικό χρονικό διάστημα για να έχουμε αξιόπιστα δεδομένα που θα μας βοηθήσουν να κρίνουμε αν πρέπει να την αναθεωρήσουμε ή όχι. Δεν επιμένουμε όμως, ε, μπορεί αυτή η αναθεώρηση να γίνει στην τριετία ή στην τετραετία. Δεν επιμένουμε. Ως προς την νοσοκομιακή και μη νοσοκομιακή περίθαλψη, συμφωνώ μαζί σας ότι υπάρχει μεγάλη ε, διαφορά στους κανόνες μεταξύ των κρατών μελών για το τι θεωρείται και τι δεν θεωρείται νοσοκομιακή περίθαλψη. Προτείνουμε οι εμπειρογνώμονες ε, των κρατών μελών ε, με τη διαδικασία της επιτροπολογίας να λάβουν αποφάσεις σχετικά με το τι θα θεωρείται και τι όχι νοσοκομιακή περίθαλψη. Αλλιώς θα έχουμε μια μεγάλη σειρά ορισμών και θα είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί η οδηγία ως προς ε, την νομική βάση και θα κλείσω. Προσωπικά θα ήθελα πάρα πολύ το άρθρο 152 ως νομική βάση. Το 152 λέει όμως το 152 μιλάει για την υγεία, δεν ε, προβλέπει όμως καμία αρμοδιότητα ε, ε, πρόθεσης νομικών μέσων. Αναφέρεται σε κίνητρα οικονομικά προγράμματα που θα βοηθούν τα κράτη-μέλη. Αναφέρεται σε συγκεκριμένα θέματα όπως είναι το αίμα, η ιστή ή τα όργανα. Αλλά εάν η νομική μας υπηρεσία μου πει ότι είναι δυνατόν να βασίσουμε την οδηγία αυτή στο άρθρο 152 ή αν μπορούμε να έχουμε διπλή νομική βάση, πολύ ευχαριστώ θα το κάνω. Θα πρέπει λοιπόν οι νομικές υπηρεσίες να με συμβουλεύσουν για το θέμα αυτό. Οι συμβουλές που έλαβα μέχρι στιγμή ήταν αυτές, αλλά θα τους ρωτήσω, διότι εγώ προσωπικά θα προτιμούσα το 152. Ε, κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να ε, πάρω άλλο από το χρόνο σας, ε, αλλά προσβλέπω στη συνέχιση της συζήτησης. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ για την πολύ σημαντική αυτή ανταλλαγή απόψεων. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 28 Ιανουαρίου, την άλλη εβδομάδα δηλαδή, στις 12 η ώρα. Στις 10 ή 11 Φεβρουαρίου θα συζητήσουμε τις τροπολογίες και θα ψηφίσουμε στις 2 Μαρτίου. Θα ψηφίσουμε το σχέδιο στις 12 Μαρτίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ καθίστε γρήγορα, πρέπει να αρχίσουμε τις ψηφοφορίες και πριν το κάνουμε αυτό πρέπει να... να ρωτήσουμε τον Μάρκομ ε, Χάρβορ ε, και τον Χωσέ Περέρα σχετικά ε, με τη διασφάλιση δημοσίων υπηρεσιών υψηλής, υψηλής ποιότητας στην Ευρώπη. Uh, Συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Πρέπει να ξεκινήσουμε. Κύριε Χάρμπορ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για τους συναδέλφους που δεν ήταν χθες εδώ το απόγευμα, συμφωνήσαμε με τον κύριο Χάσε Φερέρα να αναβάλουμε την ανταλλαγή απόψεων για τις τροπολογίες στην έκθεσή μου για το διάστημα όσους πριν τις προφορίες. Παρακαλώ λοιπόν προσέξτε μας, προσέξτε μας λίγο. Ο μόνος συνάδελφος που υπέβαλε τροπολογίες για την έκθεσή μου, νομίζω, ήταν ο κύριος Άσε Φερέρα, οπότε οι υπόλοιποι σκιώδες φαντάζομαι ήταν πολύ ικανοποιημένοι με το περιεχόμενο. Όπω έχω πει και σε προηγούμενε παρεμβάσει μου, αλλά αξίζει τον κόπο να το επαναλάβω, για το ακροατήριο που βρίσκεται ακόμα στην αίθουσα, νομίζω εδώ έχουμε ένα μέσο δημόσια πολιτική που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ακόμη επαρκώ και θα δώσει πολλαπλά ωφέλη. Βελτίωση τη ποιότητα των δημοσίων υπηρεσιών. Κρίμα που κάποιοι από αυτού που ενδιαφέρονται για τι υγειονομικέ υπηρεσίε έχουν φύγει από την αίθουσα αλλά η χρήση των νέων τεχνολογιών για την παροχή υπηρεσιών είναι ένας από τους πιο ενδιαφέροντες τομείς που θα έχει και πολύ σημαντικό αντίκτυπο για τους πολίτες και την ποιότητα. Άρα θα πρέπει να τονώσουμε την ε, σημασία αυτών των, ε, των μέσων και για τις δημόσιες ε, υπηρεσίες προ όφελο των δημόσιων αρχών. Υπάρχουν πολλέ καινοτόμε εταιρείε τι οποίε μπορούν να ανατρέξουν οι δημόσιες αρχέ για να βελτιώσουν την ποιότητα και αυτό θα αλλάξει πολύ την. θα απαιτήσει να έχουμε διαφορετική νοοτροπία βεβαίω και διαφορετικό σκεπτικό και θα χρειαστεί και κατάρτιση και εκπαίδευση για να προχωρήσει μια τέτοια πρωτοβουλία. Πάντω ε, θέλω τη στήριξη τη επιτροπή μας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με αυτή την πρόταση. Να πω ότι εδώ δεν μιλάμε για νομοθετικές αλλαγές στην ουσία, αλλά για αλλαγή στη στάση και την οτροπία των ανθρώπων. Τώρα για τις τροπολογίες, Πρόεδρε, και θα περάσω και σε αυτό. Αυτό που έκανα ήταν ότι πήρα τρει από τι τροπολογίε του κ. Χάσε Φερήρα και Τις ε, συνδύασα με δικές μου. Έχουμε λοιπόν τρεις συμβαστικέ τροπολογίες, την 1, 2 και 3, οι οποίες περιλαμβάνονται ως παράρτημα στην κατάλογο ψηφοφοριών σας. Και να πω ότι και ο κύριος Λάμστορτ, εκ μέρους των φιλελευθέρων, έχει συμπαραταχθεί με την συμβαστική τροπολογία 2. Τώρα δεν ξέρω αν θέλετε να σας τι διαβάσω για να μεταφραστούν, εάν επιμένετε. Εντάξει, δεν πειράζει. Επίσης υπάρχει και μια προφορική τροπολογία, την οποία θα σας διαβάσω μάλλον, διότι πρόκειται για ουσιαστική διευκρίνηση και καλύτερη διατύπωση του τι μπορούν να κάνουν οι προμήθειες πριν από το εμπορικό στάδιο. Και ορίζει και ένα πλαίσιο για όλη την έκθεση η τροπολογία αυτή καλωσορίζει τη διευκρίνηση της Επιτροπής ότι οι προμήθειες πριν από το εμπορικό στάδιο μπορούν να διενεργούνται από τις ε, σημαντικές αρχές τη στιγμή της έρευνας πριν από την ε, θέση σε εμπορία. Αυτό σημαίνει το σχέδιο, την καταγραφή του πρωτοτύπου, τον περιορισμένο όγκο των πρώτων προϊόντων και υπηρεσιών σε μια σειρά δοκιμών και μια τέτοια σφαιρική προσέγγιση θα διευκολύνει την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στι δημόσιε προμήθειε, κάνοντα διάκριση μεταξύ τη φάση τη καινοτομία, τη καινοτόμου έρευνα και τη θέση σε εμπορία. Είναι πολύ δύσκολο κάποιε φορέ να χρηματοδοτηθούν οι, νέες, οι νεαρές εταιρείε και ούτω καθεξής. Νομίζω, Πρόεδρε, επιφέρει διευκρίνηση η τροπολογία αυτή. Καλό θα είναι λοιπόν να στηριχθεί Κύριε Φερέρα, Χάσε Φερέρα, θέλετε το λόγο. Έχετε κάποιο σύντομο σχολείο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Η έκθεση αυτή είναι πολύ σημαντική νομίζω για να ενισχύσουμε τη διαδικασία της χειροτομίας στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Κατά τρόπο βιώσιμο και ουσιαστικό, επιτρέποντας τις δημόσιες αρχές δηλαδή, να συμπεριλάβουν τα ωφέλη από μια τέτοια διαδικασία σε προτάσεις που διατυπώνονται από εταιρείε διαφορετικών διαστάσεων και εγκυόμενες συνθήκες ε, τέτοιες ώστε οι μικρότερες επιχειρήσεις να μπορούν να αναλάβουν δράσεις στους τομείς της καινοτομίας και της έρευνας. Έτσι οι πολίτες και οι καταναλωτές θα ωφεληθούν από την όλη διαδικασία. Η έκθεση, ο κύριος ε, μάλλον ο εισηγητής με την έκθεση του, ο κύριος Μάλκομ Χάρμπορ, έχει υποβάλει ένα κείμενο που νομίζω ότι θα έχει γίνει εξαιρετικό αφού έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση για τις τροπολογίες. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων και διαπραγματεύσεων που έγιναν, μπορέσαμε να διασκεδάσουμε όλες τις ανησυχίες και τους ενδιασμούς που είχαν αναφερθεί και από μένα τον ίδιο και από τον εισηγητή. Κατά αυτόν τον τρόπο το αποτέλεσμα τελικά συμπεριλαμβάνει συμβιβαστικέ λύσεις όπως μας προείπε ο κύριος Χάρμπορ και γίνεται μια καλή επιλογή των προτάσεων για αλλαγές. Καλύπτουμε κενά του κειμένου και Τώρα πραγματικά εμβαθύνουμε στην ουσία του θέματος, γίνεται πιο ακριβές το κείμενο, πιο ευανάγνωστο και πιο λειτουργικό. Ολοκληρώνοντας, Πρόεδρε, να τονίσω ότι η θέση μου είναι σαφώς υπέρ της έγκρισης του κειμένου και υπέρ των, των περισσότερων τροπολογιών. Νομίζω πάντως ότι η Επιτροπή μας μπορεί να ολοκληρώ, να εγκρίνει συνολικά το κείμενο και στη συνέχεια το κείμενο αυτό να γίνει αποδεκτό και από το Κοινοβούλιο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστούμε. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο εφόσον χρειάζεται. Κύριε Λάσλο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την καλή δουλειά που έκανε και να πω ότι η πολιτική μου ομάδα ε, στηρίζει τις ε, δύο ε, συμβαστικές τροπολογίες, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, η προφορική τροπολογία του συναδέλφου Χάρμπορ, η οποία είναι επί της ουσίας. Ο κίνδυνος με την προφορική αυτή τροπολογία είναι, και γι' αυτό θα ήθελα να την καταψηφίσετε, είναι ότι από τη μία ε, έχουμε την ε, φάση ε, έρευνας και ανάπτυξης και από την άλλη την φάση παραγωγής και με την τροπολογία αυτή δεν γίνεται σαφής διάκριση αυτών. Ε, για παράδειγμα, στην ε, οδηγία για τον ε, τομέα ασφαλείας έχουμε ορίσει σαφώς πού τελειώνει η φάση της έρευνας, έρευνας και ανάπτυξης και πού ξεκινάει η φάση της ανάπτυξης. Εδώ πέρα λοιπόν την διάκριση αυτή την έχουμε σβήσει ουσιαστικά. Δεν είναι αρκετά σαφή η διάκριση και νομίζω ότι έτσι κάνουμε ένα επικίνδυνο άνοιγμα με την προφορική αυτή τροπολογία. Αυτό είναι το μόνο θέμα που διαφωνώ με την έκθεση αυτή κατά άλλα. Συμφωνώ πολύ με την καλή αυτή ε, έκθεση. Θα ήθελα λοιπόν να καταψηφίσετε αυτήν την συγκεκριμένη προφορική τροπολογία για να γίνει σαφή διάκριση ανάμεσα στη φάση έρευνα και ανάπτυξη και στη φάση παραγωγή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Από μπορούμε να ξεκινήσουμε να ψηφίζουμε. Παράγραφος 1. Τροπολογία μάλλον 1, λέει πρόεδρος. Τροπολογία 2. Υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται. Τροπολογία Ήτρε. Υπέρ. Κατά. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 1. Υπέρ κατά εγκρίνεται επτά υπέρ κατά εγκρίνεται οκτώ υπέρ κατά εγκρίνεται εννέα υπέρ κατά εγκρίνεται δέκα υπέρ κατά εγκρίνεται 11 υπέρ κατά εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά εγκρίνεται. 3 της Γιούρη υπέρ ευχαριστώ, κατά εγκρίνεται. 4 ευχαριστώ. 14 υπέρ ευχαριστώ κατά 2 εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά Εγκρίνεται. 15 υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 17 υπέρ. Ευχαριστώ. Α, ναι. Η προφορική τροπολογία. Κύριε Χάρμπορ. Όχι, κυρία Γκέμπχαρτ. Επιτρέψτε μου να πω κάτι γι' αυτό. Για αυτήν άκουσα το ε, επιχείρημα του κυρίου Χάρμπορ και αυτήν ε, του Γκραφ Λάμπστορφ και ε, διαπιστώνω ότι πρόκειται για μια επί της και ε, μου είναι δύσκολο να κρίνω τις ε, συνέπειε. άλλωστε την τροπολογία αυτή την έχουμε λάβει μόνο στα αγγλικά και όχι στην ε, γλώσσα εργασία μου τα γερμανικά. προτείνω λοιπόν να μην ψηφιστεί αυτή η προφορική τροπολογία. προτείνω να συναντηθώ με τον κύριο Χάρμπουρ και με τον κύριο Κραφ Λάμστορφ για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και να κρίνουμε τι συνέπειε αυτή τη τροπολογία, διότι τόσο γρήγορα δεν μπορούμε να κρίνουμε. Εάν ένα μέλο είναι κατά, θα ψηφίσουμε την παράγραφο 17. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 17 Επτά ήτρε λέει πρόεδρος. Όχι. Ένα της γιούρι. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Γιούρι 2 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 20 αποσύρεται. 9. Τη ΣΥΤΡΕ υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Και μετά ψηφίζουμε για το σχέδιο έκθεση συνολικά υπέρ. Υπέρ. Το 2008 ήταν το έτος της καινοτομίας. Σας συγχαίρω λοιπόν για την έκθεση. Εγκρίθηκε προφανώς. Κύριε Χάρμπορ, για την προφορική τροπολογία, να ζητήσω συγγνώμη από του συναδέλφου που δεν είχαμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε χθε. Έχει δίκιο η κυρία Γκέμπχαρτ που λέει ότι πρέπει να, το, χρόνο να το σκεφτούμε. Θα υπάρξει όμω τροπολογία ω την Ολομέλεια. Θα ακολουθήσω τους κανόνε για τι νομοδοτήσει ιδίας πρωτοβουλία. Πάντως, στο κύριο Λάστο, να πω ότι εάν και την αρχική μου διατύπωση ουσιαστικά διευκρινίζει αυτό που θέλουμε να δούμε. Δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για τα δικαιώματα των ερωτών και πετυχαίνει νομίζω τον επιδιωκόμενο στόχο. Διευκρινίζει με πολύ μεγαλύτερη προσοχή και ακρίβεια το κείμενο. Εδώ Έχετε δίκιο ότι ούτω ή άλλω πρόκειται για την περίπτωση των προμηθειών πριν από το στάδιο και το τι πεδίο δράση μπορούν να έχουν εδώ οι δημέσιε αρχέ. Εδώ πρέπει λοιπόν να δούμε τι ακριβώ θέλουμε να πετύχουμε και θα το συζητήσουμε γιατί η πείρα σα θα μα είναι πολύτιμη προκειμένου να εξεύρουμε την καλύτερη συμβαστική λύση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. 35 μέλη ενέκριναν την έκθεση. Περνάμε στην επόμενη έκθεση, Σάρλοτ Σέντερσελ, για την δημιουργία του, της, επαγγελματικής κάρτας, της Ευρωπαϊκής Επαγγελματικής Κάρτας για τους ε, παρέχοντες υπηρεσίες. Θέλετε να πείτε κάτι? Ναι. Πολύ σύντομα, απλώ να ευχαριστήσω όλους τους σκεώδεις εισηγητές. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία. Μιλάμε για την ποιότητα των υπηρεσιών και τα επαγγελματικά προσόντα είναι ένα θέμα που θα εξακολουθήσει να μας απασχολεί και στο μέλλον. Δεν είναι αυτό η τελευταία σελίδα της συγκεκριμένη ιστορίας. Παρ' όλα αυτά η συνεργασία μας ήταν αρμονική. Και όχι και υπήρξαν βέβαια κάποιες πολιτικές διαφωνίες ως προς το όλο θέμα, διαφορετικές τοποθετήσεις, αλλά όπως Προείπα αυτή είναι μόλι η αρχή της διαδικασίας. Οι επαγγελματίε του τομέα της υγείας, οι μηχανικοί, οι δικηγόροι είναι τομεί που ήδη θα μας απασχολήσουν. Και θα δούμε τι εξελίξει θα υπάρξουν και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους. Ναι, ήταν καλή συνεργασία. Νομίζω ότι έχουμε βρει καλές συμβαστικές λύσεις. Και αυτό που ήταν καλό με τη συνεργασία μας ήταν ότι δεν αποδυναμώθηκε η πρόταση. Βρήκαμε συνήθως το σημείο ισορροπίας μεταξύ δύο διαφορετικών ε, ε, θέσεων. Γι' αυτό την χαρακτήρισα καλή τη συνεργασία. other... Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας και για τη δουλειά σας. Να ψηφίσουμε λοιπόν παράγραφος 2, τροπολογία 4, υπέρ κατά, εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία υπαριθμών 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. συμβιβαστική τροπολογία 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές, να το ελέγξουμε. Τη 13 υπέρ κατά. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται λοιπόν. Περνάμε στη 15 υπέρ. Κατά. Κατά. Κανείς. Εγκρίνεται λοιπόν. Η 16 αποσύρθηκε. Συμβιβαστική τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Ένα είναι κατά. Ωραία. Εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Αποχές. Εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Α, συγγνώμη, αποχές. Εγκρίνεται, λέει ο πρόεδρος. 21 αποσύρθηκε, 22 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Και πιθανή τροφολική Προφορική τροπολογία στην 23. Ο κύριος Μπουσόη αντικατέστησα το should με το could και πρόσθεσα και το where appropriate. Ευχαριστούμε για το μάθημα αγγλικών. Υπέρ λοιπόν, κατά, εγκρίνεται με την προφορική τροπολογία 23. Όχι. Αιτιολογική σκέψη ε τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται λοιπόν. Αιτιολογική σκέψη G, τροπολογία 3, πρώτο τμήμα. Κατά τα ψηφοφορία, το πρώτο τμήμα λοιπόν υπέρ. Κατά. Το πρώτο τμήμα εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται λοιπόν. Τροπολογία υπεριθμών 1 στην παράθεση 7. Α, συγγνώμη, δεν θα την ψηφίσουμε αυτήν. Και τώρα ψηφίζουμε στο σχέδιο της έκθεσης ως τροποποιήθηκε. Υπέρ. Ευχαριστώ πολύ. Κατά. Εγκρίνεται. 34 υπερψήφισαν την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Να ψηφίσουμε τώρα την πρόταση της κυρίας Χέρτσκοκ για το σύστημα κοινοτικού οικολογικού συστήματος. Η κυρία Χέρτσκοκ απουσιάζει. Είχαμε μια καλή συνεργασία και μαζί με τον κύριο Λάνσβορ καταλήξαμε σε κάποιες συμβαστικές τροπολογίες και με την ε, συνδρομή της κυρίας Χέρτσκοκ. Να ψηφίσουμε λοιπόν την τροπολογία 5. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται λοιπόν. Συγγνώμη, απορρίπτεται. Τροπολογία 18 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Τροπολογία υπαριθμών 6 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται λοιπόν. 7D υπέρ. Απορρίπτεται λοιπόν. Περνάμε στην 8, τμήμα 1, υπέρ. Ευχαριστώ, κατά. Εγκρίνεται. 8, τμήμα, τμήμα 2, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 19, υπέρ. Όχι, δεν ψηφίζουμε την 19, περνάμε στην 8 τμήμα 3. Υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία παριθμών 9. Υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται προφορική τροπολογία στην 20. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 12 δι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 21 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 22 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Εδιολογικές σκέψεις, τροπολογία 1 υπέρ. Ευχαριστώ, κατά. Εγκρίνεται. 2 υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία υπερθυμών 1 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Και περνάμε στην 17 Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 23. Υπέρ. Υπέρ για την 23. Κατά. Απορρίπτεται. Παράρτημα 2. 24 υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 13 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Να ψηφίσουμε λοιπόν το σχέδιο γνωμοδότησης στο σύνολό του υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ξαναψηφίσουμε. Είστε όλοι υπέρ. Είναι τελική ψηφοφορία. Κατά. Αποχές. Καμία. Ωραία. Συγχαρητήρια. Τη συντάκτη της ε, γνωμοδότησης, εμένα και τον συνάδελφο που ε, περάσαμε στο συμβιβασμό. Να ψηφίσουμε τώρα τα προβλήματα και τις προπτικές της Ευρωπαϊκής Εφαγένειας. Η συγγήτρια, κυρία Γιώτοβα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον συνάδελφο για τις τρεις τροπολογίες του. Είμαι πολύ ικανοποιημένη με την εκδοχή της έκθεσης. Υπάρχει μόνο ένα σημείο στο οποίο είχαμε κάποια διαφωνία και αφορά στις συντάξεις. Εχθές καταλήξαμε σε μία συμβιβαστική πρόταση και θέλουμε να κάνουμε μία αλλαγή στην τροπολογία 3 και εκεί θα λέμε ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευκολύνουν ε, τα, τις συντάξεις και τα δικαιώματα των μισθωτών ε, ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά... Uh, um, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ιώτοβα και δέχομαι αυτό που λέει. Έτσι ευθυγραμμίζεται η οδηγία αυτή με τις άλλες. Προτείνω λοιπόν ε, να ε, ψηφίσουμε unblock όλες μαζί, δηλαδή τις τρεις τροπολογίες μου, ε, τις οποίες θα υπερψηφίσει η ομάδα μου. Ποιο Ποιος είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Μπορούμε να ψηφίσουμε τη γνωμοδότηση στο συνολό της. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν έχουμε. Εγκρίθηκε. 32 ε, ψήφοι. Ε, συγχαίρω τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές. Ψηφίζουμε την πρόταση. για τους μειωμένους συντελεστές φόρου θέμενη αξίας. Ε, η συγκητής είναι ο Όλε Σμιτ. Ε, θέλετε να σχολιάσετε πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές και όσους ε, παρενέβησαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής. Κατέβαλα κάθε προσπάθεια για να ακολουθήσω τις συμβουλές σας. Μία μόνο τροπολογία δεν με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο, η τροπολογία 4. Κατά τα άλλα όμως έχουμε καταλήξει σε μια πολύ ε, καλή και χρήσιμη κοινή θέση. Ευχαριστώ. Ε, τροπολογία 4, ε, διολογική σκέψη 3. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεν έχουμε. Απορρίπτεται. Ε, συμβαστική τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και μπορούμε να συμφίσουμε την έκθεση στο σύνολό Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Ευχαριστώ. Συγχαίρω τον εισηγητή. Κατόπιν έχουμε την έκθεση του κυρίου Τσίμπη για τον ενεργό διάλογο με τους πολίτες ε, σχετικά με την Ευρώπη. Κύριε Τσίμπη, δεν θέλετε να σχολιάσετε. Ωραία, μπορούμε να ψηφίσουμε. Συμβαστική τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 4. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ. Πρέπει να το ελέγξουμε. 6. Τροπολογία 6. Ε, 17 υπέρ. Ε, ποιος είναι κατά, συγγνώμη, κατά. Εγκρίθηκε. 7 υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Συμβιβαστική τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. 9 υπέρ κατά εγκρίθηκε 10 υπέρ Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά εγκρίθηκε. 13 υπέρ κατά εγκρίθηκε και τελική ψηφοφορία υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαίρω τον εισηγητή. Κατόπιν έχουμε τον ε, Επίτροπο Μακρύβη. Είναι παρόν. Σε δύο-τρία λεπτά θα συνεχίσουμε. Ο κύριος Μακρύβη έρχεται και μπορούμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας.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 Αγαπητοί συναδελφοί, και να περάσουμε στο επόμενο σημαντικό σημείο της Μερίσιας διάταξης. Έχουμε συζήτηση με τον Επίτροπο Μαγκρίβη για την αναθεώρηση της ενιαίας αγοράς. Θα ήθελα καταρχάς να σας καλωσορίσω κύριε Μαγκρίβη και να σας ευχαριστήσω που έρχεστε εδώ στην Επιτροπή μας. Να σας υπενθυμίσω ότι η Επιτροπή μας ακολούθησε την ε, αναθεώρηση της ε, αγοράς ε, στενά του 2007 και αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ε, λόγω και της παρούσας οικονομικής κατάστασης. Θα ήθελα να σας ζητήσω κύριε Μακρύβη να μας πείτε λίγα πράγματα για τις εξελίξεις που είχαμε μετά την αναθεώρηση του 2007 και τι έγινε με την ε, παρακολούθηση της ε, αγοράς λιανικών πωλήσεων. Θα ήθελα να ξέρω και κάποια πράγματα για το πώς έχει εφαρμογή τις οδηγίες για τις υπηρεσίες στα κράτη-μέλη και ε, τι γίνεται για τις οδηγίες για το scoreboard της εσωτερικής αγοράς. Θα ήθελα να σας πω ότι η Επιτροπή παρακολουθεί στενά το σύστημα Solvit και ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το πρόγραμμα ε, δράσης για τον εξορθολογισμό όλων των συστημάτων της εννέας αγοράς. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, συγχωρήστε με για τη φωνή μου. Έχω κρυολογήσει Έχω αυτή την επιδημία γρήπης που οι περισσότεροι πέρασαν θα περάσουν ή περνάνε. Και πρέπει να πω ότι εφόσον είναι πρώτη μας συνάντηση για φέτος, να ευχηθώ και καλή χρονιά και ό,τι καλύτερο για το 2009. Ίσως αυτή να είναι η τελευταία μου επίσκεψη στην Επιτροπή σας κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας. Ήθελα λοιπόν να εκφράσω την εκτίμησή μου για την εξαίρετη συνεργασία που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Καταφέραμε να προχωρήσουμε πολύ στην εσωτερική αγορά, αλλά φυσικά η δουλειά μας δεν έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχουν ε, σωματικές προκλήσεις για το άμεσο μέλλον. Είναι δύσκολες στιγμές αυτές που περνάνε οι καταναλωτές και επιχειρήσεις. Οι οικονομικές προβλέψεις είναι ε, δυστυχώς ε, σκοτεινέ, ζωφερές και συνεχώς χειροτερεύουν. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε λοιπόν πολύ μεγάλες προκλήσεις Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλη μας την επινοητικότητα και την ευθεία για να προσπαθήσουμε να βγούμε από τη σημερινή οικονομική κρίση. Για το 2009 και μετά θα πρέπει να σχεδιάσουμε μια νέα μορφή για τις πολιτικές. Και η οικονομική κρίση σαφώς δεν θα ξεπεραστεί χωρίς τα εργαλεία της εσωτερικής αγοράς. Στην εσωτερική αγορά μπορούμε να αναζητήσουμε τα στοιχεία που θα μας επιτρέψουν να ανακάμψουμε στην Ευρώπη. Μια συνολική προσπάθεια πρωτοβουλία της Κομισιόν αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη για να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε την οικονομική κρίση με νομοθεσία και ενισχύοντας την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα με ελαστικότητα και με ταχύτητα. Σε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη και την Προεδρία του Συμβουλίου και για να στηρίξουμε τις τράπεζες. Χρειαζόμαστε λοιπόν απαραίτητε προσαρμογέ στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι οποίε θα αφορούν τι κεφαλαιοχικές απαιτήσει των τραπεζών, του χρηματοπιστωτικού οργανισμού και θα πρέπει να γίνουν και να υποβληθούν όσο το δυνατόν συντομότερα. Αυτό πρέπει να το πράξουμε άμεσα, γιατί ο κίνδυνο δεν θα περάσει έτσι εύκολα. Και επίση έχουμε λάβει και τα πρώτα αποφασιστικά βήματα για να αντιμετωπίσουμε την ε, ύφεση τη πραγματική οικονομία. Το Συμβούλιο στηρίξει την πρόταση τη Επιτροπής για, για το σχέδιο οικονομική ε, ανάκαμψη τη Ευρώπη. Τα προβλήματα και τους κινδύνους που σήμερα διατρέχουμε μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε μόνο ενωμένοι. Το μήνυμά μου σήμερα για σας είναι ότι η εσωτερική μας αγορά θα είναι μέρος αυτής της προσπάθειας. Είναι ο τομέας της αρμοδιότητάς σας. Είναι η εσωτερική αγορά που πρέπει να διατηρήσουμε και να αναπτύξουμε περαιτέρω και για σήμερα και για το μέλλον. Έχουμε τόσα εκατομμύρια ανθρώπους στην εσωτερική αυτή αγορά και ένα κοινό νόμισμα που μπορεί να είναι θύματα της ύφεση και της κρίσης. Θα πρέπει λοιπόν στο μέλλον να σχεδιάσουμε το πώς θα έχουμε μια μακροπρόθεσμη ανάκαμψη. Η εσωτερική αγορά είναι σημαντική για τους καταναλωτές και τους επιχειρηματίες. Πρέπει να τους βοηθήσουμε λοιπόν να επενδύσουν και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και οι τράπεζες να δανείσουν ξανά. Η αναθεώρηση της εσωτερικής αγοράς πρέπει να συμβάλλει συγκεκριμένα στην αντιμετώπιση της κρίσης. Όπως ξέρετε πριν από μερικές εβδομάδες υπέβαλα την πρώτη ετήσια έκθεση για την αναθεώρηση, την επισκόπηση του τι έγινε στην εσωτερική αγορά το 2007. Στις 16 Δεκεμβρίου του 2008 υπευλήθη, δημοσιεύτηκε η έκθεση αυτή με αποτελέσματα και πορίσματα πολύ σαφή και ακριβή και νομίζω ότι μας οδηγεί να σκεφτούμε συγκεκριμένα θέματα που έχουν να κάνουν με την ανάκαμψη και τα οποία θα προσπαθήσω να διαγράψω εν συντομία. Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να στηρίξουμε τους πολίτες και τους καταναλωτές για να αντιμετωπιστεί η κρίση. Πολλά πράγματα έχουν επιδεινωθεί από το 2007. Η προστασία των καταναλωτών όμως και οι επιλογέ των καταναλωτών στην ελληνική αγορά είναι πράγματα που μπορούν να στηριχθούν και με βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Θέλουμε εναρμόνιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά με την πρόσφατη πρότασή μα. Θα πρέπει να έχουν το ίδιο επίπεδο προστασία παντού στην Ευρώπη οι καταναλωτέ. Και αυτή ακριβώ την πρόταση πρέπει να εξετάσει και η Επιτροπή σα. Στον τομέα των, ε, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, των αποταμιεύσεων, των τραπεζικών υπηρεσιών, ε, θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προτεραιότητα. Και ήδη αυτό έγινε το 2008. Ήδη είχαμε συμφωνία με τον τραπεζικό κλάδο για το πώς θα συνεργάζονται οι τράπεζες μεταξύ τους και για επενδυτικά προϊόντα που θα διατεθούν σύντομα στους καταναλωτές, ώστε να αυξηθεί η εμπιστοσύνη τους και το επίπεδο προστασία τους. Είναι πολλά τα ανταγωνιστικά επενδυτικά προϊόντα από τα οποία θα μπορούν να διαλέξουν. Μόνο οι καλά ενημερωμένοι πολίτες και καταναλωτές μπορούν να κάνουν και σωστές επιλογές. Γι' αυτό ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα όπου η εσωτερική αγορά θα περιλαμβάνει νέες υπηρεσίες και μια κοινή ε, δίωδο ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που μπορεί αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίζονται με την έλλειψη καταμόνησης στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες θα φροντίζουμε να ενημερώνουμε σταθερά και συστηματικά την Επιτροπή σα για τι εξελίξει στον τομέα αυτό. Επίση, η εσωτερική αγορά μπορεί να καλύψει τα συμφέροντα των μικρών επιχειρήσεων που παίζουν ζωτικό ρόλο σε ό,τι αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασία. Προτεραιότητά μα για το 2009 είναι να εγκριθεί ένα υγιέ περιβάλλον, κυρίω για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Πολλέ προτάσει μεταρρύθμιση ε, εξετάζονται αυτή τη στιγμή από το Συμβούλιο Ιδίω για το πώ μπορούμε γρήγορα να διαθέσουμε ποσά στι μικρέ υπηρεσίε. Επίση υπάρχει πρόταση του περασμένου Ιουνίου για, το ενιαίο και απλουστευμένο καθεστώ των μικρών επιχειρήσεων. Εδώ χρειάζεται να γίνει μια σημαντική διάκριση ώστε να έχουν και τα κράτη-μέλη την δυνατότητα να ε, εξαιρέσουν μικρές επιχειρήσεις από τους κανόνες για τα λογιστικά πρότυπα. Εδώ η ταχύτητα θα είναι ζωτικής σημασίας θα πρέπει τα κράτη-μέλη να αφήσουν κατά μέρο του ε, εθνικού ενδιασμού και τα δικά του ε, ειδικά συμφέροντα για να φτάσουμε σε συμφωνία. Γιατί οποιαδήποτε τέτοια πρόταση μα οδηγήσει σε ενοποίηση του συστήματο θα είναι ευπρόσδεκτη. Επίση υπάρχουν και άλλε προκλήσει που έχουν να κάνουν με την ουστική αγορά και σχετίζονται και με την ενδεχόμενη ανάκαμψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή θέλει να φροντίσει οι αρχές που διέπουν την εσωτερική αγορά να εφαρμόζονται σωστά και να υπάρχει ένα ε, να υπάρχει ισοτιμία στον ανταγωνισμό μεταξύ όλων. Αυτή η ισοτιμία στον ανταγωνισμό θα είναι ακριβώ και η θεμέλιο λήθο για την ε, περαιτέρω ανάπτυξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτι στο οποίο βασιστήκαμε εδώ και δεκαετίε. Αν δεν είχαμε δημιουργήσει την εσωτερική αγορά, είμαι βέβαιο ότι θα έπρεπε για να αποκριθούμε στη σημερινή κρίση να τη δημιουργήσουμε ούτω ή άλλω. Θα πρέπει βεβαίω να αναλάβουμε και συγκεκριμένε δράσει σε πολλού τομεί πολιτικού τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή θα συνδράμει και θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη όπου χρειάζεται. Στο δικό μου τομέα λόγω χάρη θα πρέπει να εφαρμόσουμε μια πολιτική επιταχυμένη για τι δημόσιες προμήθειε από το 2009-2010 με συγκεκριμένα προϊόντα. Επίση, θα συνδράμουμε τα κράτη-μέλη αναλαμβάνοντα εθνικά προγράμματα αποκατάστασης για να βρεθούν λύσεις σε περιπτώσεις προμηθειών. Η αναθεώρηση της εσωτερικής αγοράς σκοπό έχει να διευρύνει την εταιρική μας σχέση με τα κράτη-μέλη σε όλους τους πολιτικούς κλάδους. Τον Ιούνιο πρόκειται να παρουσιάσω μια σύσταση τη Επιτροπή για την κοινή διαχείριση τη εσωτερική αγορά. Η σύσταση αυτή θα λαμβάνει μια σειρά δράσεων που μπορούν να αναλάβουν τα κράτη-μέλη προκειμένου να μεταφέρουν, να υλοποιήσουν και να επιβάλλουν του κανόνε τη εσωτερική αγορά και με τρόπου που να πληροφορούν καλύτερα του πολίτε για τα δικαιώματα που του ε, δίνει η εσωτερική αγορά. Για να δούμε πώ μπορούμε να βελτιώσουμε την εγχώρια αλλά και τη διασυνοριακή συνεργασία στα κράτη-μέλη. Επιπλέον, για να τονώσουμε τη διαδικασία αυτή, θα πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει και με την ποιότητα τη ε, μεταφορά, καθώς και με τον πίνακα βαθμολογίας της αγοράς. Θα δούμε πώς, ε, ε, τι επίδοση έχουν τα κράτη-μέλη σε σχέση με τις παραβάσεις, ποια, τι κάνουν με τους οικονομικούς δείκτες και τι επιτυχία μπορεί να έχουν. Τέλος, θέλω να μιλήσουμε για την πρόοδο στην εφαρμογή της οδηγίας περιπηρεσιών. Η συλλογιστική μας μας έχει να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο και μια ενοποιημένη διαδικασία αμοιβαίας ε, αξιολόγησης. Κάναμε μια, αποτίμη, μια, αξιολόγη, μια εκτίμηση του τι έκαναν τα κράτη-μέλη στην εσωτερική αγορά τα, τον τελευταίο χρόνο. Και είδαμε ότι τα κράτη-μέλη σε τομείς προτεραιότητας έχουν αποδώσει τα κονδύλια που απαιτούνταν. θα πρέπει να αυξήσουμε εδώ τις προσπάθειές μας. Τα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή προβλέπουν ε, πρακτικές συγκεκριμένες λύσεις για το σημείο επαφής, το ενιαίο σημείο επαφής και καταβάλουν και τα απαραίτητα κονδύλια. Επίσης, οι ηλεκτρονικές διαδικασίες θα επιτρέψουν στους παρέχοντες υπηρεσίες να χρησιμοποιήσουν τέτοια μέσα απλοποιημένα προκειμένου να προσφέρουν τα προϊόντα τους. Οι... Τα κράτη-μέλη προσπαθούν να θεωρήσουν την νομοθεσία τους και, την νομοθεσία τους και αυτό θα πρέπει να το κάνουν στο δυνατόν συντομότερα. Η διαδικασία αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί με ταχύτητα ώστε τα κράτη-μέλη να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα νομοθετικά μέτρα εγκαίρως. Και θα πρέπει να υποβάλουν και έκθεση μέχρι την προθεσμία για την ε, μεταφορά και μέσω της ε, διαδικασίας ε, αξιολόγησης να αποτιμηθεί η προσπάθειά τους και συμβολή τους στην εσωτερική αγορά. Αυτή είναι μια λεπτομερής εικόνα του πού βρισκόμαστε σε σχέση με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά θα ενημερώνουμε διαρκώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις εξελίξεις σε όλη αυτή τη διαδικασία. Επίσης θα πρέπει να αναλάβουμε πρακτικές διαθετήσεις για την διοικητική συνεργασία μεταξύ των τοπικών ε, αρχών. Υπάρχει ένα πιλωτικό σχέδιο σε σχέση με την οδηγία των υπηρεσιών και τα κράτη-μέλη βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη διαδικασία του εντοπισμού των ε, αρμόδιων αρχών που θα αναλάβουν Έπειτα, μετά, τη φάση των, μετά από την καταγραφή των αρχών αυτών, θα περάσουμε στη φάση των δοκιμών. Για όλα αυτά είναι ζωτική σημασία στα κάτι μελη να αποδώσουν του απαραίτητου πόρου στην ευαισθητοποίηση του κοινού και στην κατάρτιση των μελλοντικών χρηστών του συστήματο, αυτού πληροφόρηση για την εσωτερική αγορά. Και η Επιτροπή βέβαια θα παρέσχει τεχνική συνδρομή, θα παρακολουθεί, θα διευκολύνει και θα συντονίζει όλο αυτό το έργο. Αυτέ τι προκλήσει μπορούμε να τι αντιμετωπίσουμε και να πετύχουμε του στόχου μα μόνο αν τα κράτη-μέλη αποδώσουν του απαραίτητου πόρου και καταβάλουν όσε δυνατέ προσπάθειε. Εγώ θα φροντίζω να σα ενημερώνω διαρκώ για τη διαδικασία υλοποίηση και για το πώ πηγαίνει η διαδικασία αξιολόγηση. Θα ζητήσω λοιπόν και την πολιτική σα στήριξη καθώ και την άσκηση πίεση στα κράτη-μέλη για όλα αυτά τα θέματα. Συνολικά, η εσωτερική αγορά μπορεί να χρησιμεύσει ω μέσο για την αντιμετώπιση τη ανάκαμψη. Πρέπει να διασώσουμε θέσει εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά κύριο λόγο. Η, υπηρεσία, η οδηγία των υπηρεσιών είναι ένα καλό μέσο για να δημιουργηθούν νέε θέσει εργασία και για οικονομική ανάπτυξη μέσα στο πλαίσιο τη σημερινή ύφεση. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να καταβάλουμε προσπάθειες για αυτό. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα, όταν μιλάμε για τις μεμονωμένες πτυχές ε, της ενιαίας αγοράς και όταν κοιτάμε τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής ε, στην Επιτροπή μας, ε, βλέπουμε ότι κατά τη θητεία μας διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μεγάλο κενό στο ηλεκτρονικό εμπόριο στην ε, οδηγία για την εμπιστοσύνη του καταναλωτή στο ψηφιακό περιβάλλον. Λέμε ότι μπορούμε να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη αυτή αν ορίσουμε σαφώς ε, τους κανόνες ε, και τα δικαιώματα των καταναλωτών και να ενημερώσουμε τους καταναλωτές για τα δικαιώματά τους. Είπαμε ότι χρειαζόμαστε συγκεκριμένα μέσα ώστε η Ευρώπη να μπορεί να γίνει ανταγωνιστική και στο θέμα εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Μία από τις προτάσεις ήταν να δίνονται πληροφορίες ε, στους καταναλωτές για τα δικαιώματά τους ε, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στο εμπόριο μέσω διαδικτύου. Η Επίτροπος Κούνεβα συνέταξε οδηγίες χρηστών που ε, πρόκειται να δημοσιευτούν το καλοκαίρι στο, στην ιστοσελίδα της ε, Κομισιόν. Ε, λείπει όμως κάτι εδώ ε, ό,τι αφορά την διανοητική ιδιοκτησία και αυτό είναι κάτι ε, που αφορά τη δική σας γενική διεύθυνση. Μπορείτε σας παρακαλώ να βεβαιωθείτε να ολοκληρωθεί το θέμα αυτό διότι θέλουμε μέχρι το τέλος της θητείας μας να είναι διαθέσιμη στην ιστοθέση της, να διαθέσιμος στην σελίδα της Κομισιόν ο οδηγός Χριστών αυτός. μια έκκληση για σας δηλαδή. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στους συντονιστές καταρχήν στον κύριο Χάρμπορ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν Θα ήθελα να επενέσω τον Τσάρλι Μακρύβη για την πολλή δουλειά που έχει κάνει για να προωθήσει την ενιαία αγορά και για τον ενθουσιασμό του ε, όσο καιρό βρίσκεται εδώ μαζί μας. Ε, απογοητεύτηκα που άκουσε ότι ε, η σημερινή είναι η τελευταία του παρουσία στην Επιτροπή μας. Ε, ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε στο πρόγραμμά μας μια μέρα να τον ξαναδούμε, να τον αποχαιρετήσουμε σωστά, ε, να πιούμε και κάτι μετά ενδεχομένως. Ε, ο συνάδελφος συμφωνεί. Υπάρχει μια σειρά επιτευγμάτων, εκ των οποίων η οδηγία για τις υπηρεσίες ε, ήταν η σημαντικότερη, διότι η αγορά υπηρεσιών που εκτιμάται ότι ε, αποτελεί το 70% της ευρωπαϊκής ε, οικονομίας και που πιστεύω ότι θα αυξηθεί σημαντικά ως αποτέλεσμα της παρούσας ύφεσης, ε, κάτι που λυπάμαι που το λέω, αλλά νομίζω ότι έτσι θα είναι. Αυτή η οδηγία λοιπόν είναι κεντρική σημασία και πιστεύω ότι ο συντονισμός του Επιτρόπου των Εργασιών μαζί με τη δική μας υποστήριξη έχει θέσει το πύχη και για επόμενη ε, τέτοια εγχειρήματα και η Επιτροπή μας θα πρέπει και στο μέλλον να συνεχίσει να παρακολουθεί ε, την κατάσταση στην ενιαία αγορά. Έχουν ε, επιτευχθεί ε, πολλά και πιστεύω ότι η οδηγία, η συγκεκριμένη οδηγία βασίστηκε σε όλη αυτή τη δουλειά που έχει γίνει. Πρώτη μου ερώτηση, η οποία είναι πολύ γενική. Αναρωτιέμαι μήπως ε, μπορεί ο Επίτροπος ε, με το χαρακτηριστικό του ύφος ε, να μας δώσει κάποιες, να μας κάνει κάποιες ειλικρινές παρατηρήσεις, παρατηρήσεις, να μας πει ποια είναι η θέση του. Πιστεύει ότι τα κράτη-μέλη αρχίζουν και αυτά να θέλουν να κάνουν την ενιαία αγορά να λειτουργεί σωστά. Νομίζω ότι ε, στην οδηγία κεντρική θέση ε, είχε ε, η δημιουργία στα κράτη-μέλη ενιαία θηρίδας για τις επιχειρήσεις στις χώρες τους. Με άλλα λόγια, να τεθεί πολιτικός στόχος ο οποίο δείχνει ότι η συμμετοχή των επιχειρήσεων στην ενιαία αγορά είναι κάτι καλό για τι χώρε και τις οικονομίες τους. Ε, νομίζω ότι βλέπουμε μια αλλαγή τρόπου σκέψη και σε συνδυασμό με αυτά που έκανε ο κύριο Φερχόγεν για το πακέτο για τα αγαθά. Ε, αυτά είναι δύο σημαντικά επιτέματα και θα πρέπει να τα προωθήσουμε μαζί, να τα αναφέρουμε μαζί. Η δεύτερη παρατήρηση έχει να κάνει με έναν τομέα όπου δεν πιστεύω ότι έχουμε κάνει πολύ πρόοδο. Επειδή υπήρχε ήδη νομοθεσία. Κατά τη γνώμη μου όμως ε, δεν επωφελούμαστε από αυτήν ε, όσο πρέπει και αναφέρομαι στον τομέα των δημόσιων προμηθειών. Υπάρχουν κάποιες σημαντικές ανησυχίες για τις ασυνέπειες ε, που διαπιστώνονται στις δημόσιες προμήθειες στην ενιαία αγορά. Ιδιαίτερα με απασχολεί και θα ήθελα να ακούσω αν ο Επίτροπος συμφωνεί μαζί μου και τι πιστεύει ότι μπορεί να γίνει. εμένα λοιπόν με ανησυχεί, ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι μικρές επιχειρήσεις ε, αδικούνται στις ε, δημόσιες ε, προμήθειες διότι οι δημόσιες αρχές προσπαθούν να εξοικονομήσουν χρήματα ομαδοποιώντας συμβάσεις προμηθειών και δεν συνεργάζονται με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να τις ενθαρρύνουν να υποβάλουν προσφορές. Τουναντίον οι διαδικασίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα επαχθείς και αυτό αναφέρεται στο έγγραφο για την αναθεώρηση της κοινή αγοράς. Και αναρωτιέμαι μήπως ε, ο Πίτροπο ως τελευταίο έργο πριν την αποχώρησή του ε, μπορέσει να ενθαρρύνει τις υπηρεσίες να ασχοληθούν με το θέμα αυτό, διότι στα πλαίσια της πράξη για τι μικρομεσαίε επιχειρήσεις ε, και και σε σχέση και με την αναθεώρηση τη ενιαία αγορά, ε, το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα ζωτική σημασία. Αναρωτιέμαι λοιπόν μήπω μπορεί να μα αφήσει ένα ένα φάκελο με το θέμα αυτό για να βελτιωθεί ε, το θέμα των δημοσίων προμηθειών ε, σε συνδυασμό με το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μήπω είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να αφήσει στο διάδοχό του και να το αφήσουμε εμεί στο επόμενο κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Μάντες. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συμφωνώ απόλυτα με ε, τον Μάλκολ. Πιστεύω ότι θα πρέπει να οργανώσουμε μια δεξίωση όχι για να γιορτάσουμε αλλά για να αποχαιρετήσουμε αξιοπρεπώς ε, τον Επίτροπο. Ε, χάρηκα πολύ με τη συνεργασία μας και πιστεύουμε ότι έχουμε πετύχει πολλά όπως ήδη είπε ο Μάλκολ. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Στην ε, παρουσίαση που σχετικά με την παρουσίαση που κάνατε σήμερα. Στηρίζω όλες τις προσπάθειες ε, της Κομισιόν και του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου για την, ε, ε, σχετικά με την οικονομική κρίση. Αλλά θέλω να ξέρω τι κάνουμε για τους καταναλωτές, από τι, τι κάνουμε από την πλευρά της συζήτηση, Για παράδειγμα, για την αυτοκινητοβιομηχανία. Ε, στην αυτοκινητοβιομηχανία δίνουμε εύκολα δάνεια αλλά εάν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μπορέσουμε να εισάγουμε μέτρα δημοσιονομικά σχετικά με την αγορά νέων αυτοκινήτων από τους καταναλωτές. Αυτό είναι ε, ε, επένδυση αφενός στην αυτοκινητοβιομηχανία, αφετέρου ε, για να αλλάξει το όλο κλίμα. Αυτό θα ήταν καλό για όλους. Το άλλο που θα ήθελα να γνωρίζω είναι πότε μπορούμε να περιμένουμε, μπορεί να μου πείτε ποτέ, πότε μπορούμε να περιμένουμε την οδηγία για το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνία για να μπορέσουμε πράγματι να προστατεύσουμε τις καινοτόμε ιδέε μας, εφευρέσεις κλπ. Φέτος, όπως θα γνωρίζετε, το 2009 είναι το έτος της καινοτομία και της δημιουργικότητα. Και μια τελευταία παρατήρηση, σαν πρόταση που ενδεχομένω να την υποβάλλετε. Μια ιδέα για την, στην οικονομική μας κρίση. Οι κυρώσεις που τα πρόστιμα που μαζεύει η συνάδελφό σας η κυρία Κρού, να ε, επανισχωρούν στη βιομηχανία στηρίζοντα ε, νέε καινοτόμε επιχειρήσει αντί να μειώνεται η συμβολή των κρατών μελών. Ε, ευχαριστώ πολύ. σα ευχαριστώ για τη συνεργασία τα τελευταία πέντε χρόνια και ελπίζω να μπορέσουμε αργότερα να φύγουμε από ποτό μαζί. Ο κύριος Σουάπ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Στην εισαγωγή σας ήδη είπατε ότι προφανώς για τελευταία φορά εμφανίζεστε εδώ στην Επιτροπή μας ως Επίτροπος ε, και ότι είναι η τελευταία φορά που μας μιλάτε για την ε, σχετική σας δουλειά. Ε, πριν τη σημερινή συνεδρία, κάσα και έψαξα τα ε, τελευταία πράγματα που έχετε δημοσιεύσει και μου έκανε εντύπωση ότι λέτε στην αναθεώρηση της, κοινο... της ε, κοινή αγοράς ότι πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση ε, και στα, ε, στο Κοινοβούλιο, το Κομισιό του Συμβούλιο, αλλά και στα κράτη-μέλη. Και σας ρωτώ, είσαστε πεπισμένος ότι τα κράτη-μέλη είναι έτοιμα να συνεργαστούν πιο στενά μαζί με την ε, Κομισιόν, μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή πιστεύετε ότι έχει επιδεινωθεί η συνεργασία. Η ε, οδηγία για τις ε, υπηρεσίες, η οδηγία για την πληροφόρηση των ασθενών, ε, μας δείχνουν το αντίθετο. Έχουμε το Βάξλα Κλάους στη, στη Τσεχία, ε, στην Ιρλανδία ε, έχουμε επίσης προβλήματα. Πιστεύετε λοιπόν ότι οι, πολίτες είναι, οι χώρες είναι όντως έτοιμες να συνεργαστούν καλύτερα με ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ε, αντιλαμβάνονται οι πολίτες την ενιαία αγορά ως ευκαιρία. θα ήθελα λοιπόν να ακούσω τις παρατηρήσεις σας τώρα στο τέλος της θητείας σας. Και το, η δεύτερη μου παρατήρηση είναι αυτή της, του, ενιαίου του Ευρωπαϊκού Χώρου Ενιαίων Πληρωμών. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ε, ενιαίας αγοράς και έχει να κάνει με τις ε, πληρωμές μέσω τραπεζών κλπ. Ε, δεν υπάρχει νομίζω σαφές ε, χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να ε, εκπονηθεί ε, ένα ενιαίο έντυπο. Τι πρέπει να γίνει για να εφαρμοστεί αυτό μέχρι το τέλος της χρονιάς, διότι υποτίθεται ότι θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου του 2010. Και η τελευταία μου παρατήρηση είναι ότι στο παρελθόν έχετε αναλάβει πρωτοβουλίες για την ε, ενιαία αγορά, ιδιαίτερα ως προς την ε, ανάθεση συμβάσεων. Έχουμε συζητήσει ε, το θέμα αυτό, έχουμε ψηφίσει την έκθεση για τις προμήθειες στον αμυντικό τομέα, είχαμε και άλλα σχετικά νομοθετήματα. Η ευελιξία αυτή λοιπόν ε, ε, όντως είναι κάτι που μπορεί να μας ε, ωφελήσει. Θα παρακαλούσα να μας σχολιάσετε το θέμα αυτό και θα χαρώ κι εγώ πάρα πολύ αν μπορέσουμε να πιούμε μια πίρα μαζί. Ευχαριστώ. Irish beer, yes. Ιρλανδική μπύρα, ναι. Κόρντα. Η κυρία Κόρντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, είναι πολύ άριθμα τα παραδείγματα που μας επισημαίνουν οι πολίτες μας καθημερινά καθώς και διάφορες οργανώσεις οι οποίοι μας μιλούν για τους φραγμούς που εμποδίζουν την υλοποίηση, την πραγματοποίηση της ε, εσωτερικής αγοράς. Να σας δώσω δύο πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα άρνηση κάποιων εταιριών που έχουν έδρα σε ένα συγκεκριμένο κράτος και πολλούν ε, με ταχυδρομικά ε, αρνούνται να παραδώσουν τα προϊόντα τους σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία και σας δίνουν τη διεύθυνση που τους βολεύει. Βέλγιο και Γαλλία λόγου χάρη. Αντιλαμβάνομαι ότι κάποια προϊόντα στη Γαλλία μπορεί να είναι πιο φτηνά, τα ζητάω στη Γαλλία και θα πρέπει και αυτό που θα συμβεί είναι ότι με παραπέμπουν στην έδρα της ίδιας εταιρεία στο Βέλγιο. Αν μιλάμε για ενιαία αγορά και εσωτερική αγορά, αυτό δεν επιτρέπεται. Ή μετά εκδότες κάποιων πιστοτικών καρτών, οι οποίοι αρνούνται τη χρήση κάποιων καρτών. Ξεκινώντας είπατε ότι πρέπει να περάσουμε από, να ξεπεράσουμε τέτοιου είδους φραγμούς. Δεν μπορούμε τέτοια προβλήματα, τέτοιες, τέτοια εμπόδια της ελεύθερης κυκλοφορίας να τα αγνοούμε. Πώς θα αντιδράσετε λοιπόν για να οδεύσουμε σε αυτή την αγορά που όλοι ελπίζουμε να έχουμε κάποια στιγμή, την οποία προσδοκούν όλοι οι πολίτες. Άλλες ερωτήσεις. Ο κύριος Ροζεφερέρα. you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, σας ευχαριστούμε για το λόγο που εκφωνήσατε εδώ σήμερα. Ήταν αποφασιστικός ο ρόλος σας στην έγκριση αυτής της οδηγίας. και άλλοι συνάδελφοι όπως ο κύριος και η κυρία θυμούνται ότι τα συζητήσαμε αυτά και εντατικά και με ισχυρές απόψεις. Το ενδιαφέρον για αυτή τη διαδικασία είναι όλο ένα αυξανόμενο σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπου ετοιμάζεται με διαφορετικούς ρυθμούς κατά τις πληροφορίες μου και διαδικασία μεταφοράς. Δεν ξέρω αν θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποια συνοπτική εικόνα για το πώς προχωράει αυτή η διαδικασία. Πώς προετοιμάζονται για τη μεταφορά οι διάφορες χώρες. Πώς εξελίσσεται η μεταφορά. Όταν το συζητήσαμε αυτό εδώ, νομίζω ότι καταλήξαμε ότι όλοι στην Ευρώπη γνωρίζουμε από την πρώτη φάση της συζήτηση για την οδηγία Μπόλκενστάιν ότι η οδηγία αυτή, τα μέτρα αυτά προέρχονται από την Ευρώπη. Όλοι συνεργαστήκαμε για τον ίδιο σκοπό και εσείς και ο κύριος Χάρμπορ και όλοι εμείς. Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο η μεταφορά. Ένα ερώτημα λοιπόν, πώς αξιολογείται τον αντίκτυπο της ε, χρηματοπιστωτικής κρίσης στην αγορά υπηρεσιών ιδίω που συμπίπτει με την περίοδο μεταφοράς της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Τι σκέφτεστε να κάνετε. Φαντάζομαι στο Δουβλίνο σας περιμένουν διακαώς ε, συμπολίτες σας για να αντιμετωπίσετε την ε, οικονομική κρίση. Και αλλού στην Ευρώπη, κι άλλοι είναι αυτοί που θα μπορούσαν να είχαν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν. Και ιδίω αυτή η ομάδα Ιρλανδών, που δεν είναι και τόσο μικρή φυσικά, έχει ένα καθοριστικό ρόλο στη συνθήκη της Λισαβόνας και στην έγκρισή τη. Πώς θα μπορούσατε λοιπόν να συμβάλλετε στην επίλυση τέτοιων προβλημάτων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Η κυρία Πλαστίνσκα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, Έχω και εγώ την ίδια φωνή με εσάς σήμερα, την ίδια βραχνάδα. Είναι πολύ δύσκολο να πιστέψουμε ότι πέρασαν 20 χρόνια τόσο γρήγορα. Την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε θεωρούσαμε ότι θα είχε περάσει μια αιωνιότητα μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Τώρα πλησιάζει το τέλος της θητείας μας και φαίνεται ότι το ενιαίο νόμισμα τουλάχιστον ε, σε περίοδους κρίσης είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μέσο για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από την κρίση. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα που η Σλοβακία είναι το 16ο μέλος της Ευρωζώνης πλέον. Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης είναι όλο ένα και πιο ε, προφανής φέτος. Πολλές επιχειρήσεις ε, μειώνουν το προσωπικό τους και ουσιαστικά η φετινή χρονιά θα αποτελέσει μια δοκιμή για να δούμε κατά πόσον ε, η Επιτροπή μας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να είναι επιτυχή στην πράξη. Η συνεργασία μαζί σας, ε, κύριε Επίτροπε, ήταν ιδιαίτερα επικοδομητική και πέρασε πολύ σημαντική νομοθεσία κατά τη θητεία σας και θα πρέπει να δούμε τώρα τι γίνεται στην πρακτική τους εφαρμογή. Οι ηλεκτρονικές διαδικασίες ε, κρατικών προμηθειών δεν είναι τόσο καλές όσο ελπίζαμε και θα πρέπει να το προσέξουμε το θέμα αυτό. Εγώ προσπάθησα να δω πώς λειτουργεί το θέμα της μίας και μειώνης θηρίδας ε, στη Σλοβακία. Έχει ήδη ε, τεθεί σε λειτουργία το σύστημα, αλλά εξακολουθεί να έχει αρκετές εκκρεμότητες, πράγματα που πρέπει να επιληθούν. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει λοιπόν με το benchmarking και σε διάφορες περιοχές για από εκεί και πέρα να έχουμε ένα καλό πρακτικό σύστημα για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτή την οδηγία κάπως καλύτερα. Όπως είπε και ο συνάδελφος, οι δημόσιες προμήθειες ε, αποτελούν μειονέκτημα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εγώ είμαι πεπισμένη γι' αυτό. Θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν μία δημοσκόπηση για να δούμε πόσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις όντως ε, λαμβάνουν ε, δημόσιες συμβάσεις. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται σε θέματα δημοσίων προμηθειών και άμα δείτε τα πράγματα στις χώρες στις οποίες εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 οι κρατικές προμήθειες χρησιμοποιούνται ε, μόνο σε μεγάλα κονσόρσιουμ και αν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν δημιουργήσουν κονσόρσιουμ δεν μπορούν να ε, ενταχθούν καν στο διαγωνισμό. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, η κυρία Βάιλερ. Κυρία Επίτροπε, δεν θέλω να επαναλάβω ερωτήσεις που ήδη τέθηκαν, θέλω να επικεντρωθώ σε κάποια συγκεκριμένα θέματα. Πιστεύω όμως και εγώ ότι επειδή ε, πρόκειται για την τελευταία φάση της ε, συνεργασίας ε, μας μαζί σας, θα ήθελα να ακούσω τις εμπειρίες σας, όπως και ο κύριος Σβάμπ. Πώς λέει, πιστεύετε ότι θα προχωρήσει το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο στην Ιρλανδία, αλλά γενικά. Έχουμε κάνει πολλή δουλειά, ξεχάσατε ένα πολύ σημαντικό πακέτο, το πακέτο των αγαθών. Θα ήθελα πολύ ε, να μου πείτε το εξή. Ε, Νέε πρωτοβουλίε δεν θα αναλάβατε. Ε, κάτι τέτοιο πράγματι θα ήταν ανόητο, διότι σχεδόν έχουμε μπει στην προεκλογική περίοδο. Αλλά μιλήσατε για ένα νέο scoreboard, για ένα νέο πίνακα αποτελεσμάτων, για ανάλυση της παρούσας κατάστασης. σχεδιάζετε κάποιες διαδικασίες κατά κάποιων κρατών μελών ε, επειδή έχετε ήδη στην παρούσα φάση διαπιστώσει ότι κάποια κράτη-μέλη δεν έχουν εφαρμόσει σωστά ή δεν έχουν εφαρμόσει καθόλου κάποιες ε, οδηγίες ή κανονισμούς. Δεύτερον, ως προς την ανάθεση συμβάσεων πιστεύετε ότι χρειάζονται διορθώσεις ε, στη σχετική νομοθεσία με βάση τις εμπειρίες σας. Υπάρχει το κατόφλι των 5 ε, ε, εκατομμυρίων ε, και αντιστοίχω των 200.000 πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξουν τα κατόφλια αυτά. Και επίσης είπατε ότι λόγω της παρούσας οικονομικής ε, κρίσης ε, σκοπεύετε να συνεργαστείτε με την Τσεχική Προεδρία, ε, τη Γαλλία κλπ. Πώς έχουν τα πράγματα με τη συνεργασία σας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Χωρίς στενή συνεργασία δεν θα τα καταφέρουμε. Όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο δηλαδή, αλλά σε διεθνές επίπεδο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Και να, ευχαρισ... σας ευχαριστήσω εκ μέρους της ομάδας μας. Ε, δεν είχαμε πάντα αλιακάδα στη συνεργασία μας μαζί σας, αλλά γενικά... Νομίζω ότι έχουμε στηρίξει επικοδομητικά τις πρωτοβουλίες σας. Ευχαριστώ. Η Σαρλότα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Περισσότερη λιακάδα Έχουμε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω λοιπόν για την αγαστή συνεργασία και ελπίζω να μπορέσω να σας ε, αποχαιρετήσω κάπου πιο χαλαρά, όχι εδώ εδώ στην συνεδρίαση. Όταν ήρθατε είχατε ένα διεθνή αέρα, το ένιωσα και εγώ, το ένιωσαν και πολλοί άλλοι. Τώρα ε, πια αναρωτιέμαι μήπως είστε πλέον ένας από τους πιο προσγειωμένους. Παρόλα αυτά, καταφέρετε να συνεισφέρετε ουσιαστικά στην οδηγία για τις υπηρεσίες και σας είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Έχω την εντύπωση όμως ότι πλέον η ευρωπαϊκή κινητήριος δύναμη φαίνεται να έχει χάσει λίγο κάπου το σθένος της και ποιος άλλος θα μπορούσε να ανατρέψει αυτή την κατάσταση από εσάς που είσαστε εκεί από την αρχή. Πώς βλέπετε εσείς το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την εξέλιξή μας. Θεωρείτε για παράδειγμα ότι η ευρωπαϊκή οικονομική κρίση θα αναστρέψει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ή θα την πάει πίσω. Πώς βλέπετε εσείς λοιπόν τα πράγματα στο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Να θέσω κι εγώ μια ερώτηση. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Πιστεύετε ότι τα νέα κράτη-μέλη διαδραματίζουν τον πιο σημαντικό ρόλο για την προαγωγή της εσωτερικής αγοράς ή όχι. Ευχαριστώ πολύ όλα τα μέλη για τις ευχές τους. Περιμένω λοιπόν αυτή την ευκαιρία να βρεθούμε ένα βράδυ όλοι μαζί και να αποχαιρετιστούμε. Και για όσους θα μείνουν στη κοινοβούλιο και μετά τις εκλογές τους εύχομαι ότι καλύτερο. Η πρόεδρος αναφέρθηκε στα δικαιώματα για το e-commerce και το τι έκανε συνάδελφος ε, Κούνεβα και θέλατε να περάσουμε και τα θέματα των πνευματικών δικαιωμάτων ε, θα δω τι πράγματα υπάρχουν εκεί, θα δω τι μπορεί να γίνει και θα δω και τι προτάσεις υπάρχουν. Ε, θα το διερευνήσω με τις υπηρεσίες μου. Ο Μάλκον Χάρμπον έχει σε κάποια θέματα. Η οδηγία για τις υπηρεσίες ήταν το μεγάλο σου ξέρω όταν έγινα εγώ επίτροπος. Έγινα μέλος το 2004 και κυριαρχούσε πραγματικά η οδηγία για τις υπηρεσίες. κληρονόμησα μία ιδιαίτερα διαφιλονικούμενη πρωτοβουλία και η προσέγγιση που ακολούθησα μπορεί να ήταν διαφορετική από αυτή που είχαν συνηθίσει οι υπηρεσίες της Κομισιόν αλλά η προσέγγιση που υιοθέτησα βασιζόταν στην πολιτική μου πείρα και ε, την υποστήριξε και η Σάρλοτ Σίτζερχολ στο τέλος. Εγώ είμαι ρεαλιστής, είμαι πραγματιστής και αποφάσισα ότι αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε μια οδηγία για τις υπηρεσίες πρέπει να είμαστε πρακτικοί στην προσέγγισή μας. Και ρώτησα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι άλλωστε είναι και το αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας συναπόφασης και τους ζήτησα να διαδραματίσουν και αυτοί το ρόλο τους. η οδηγία για τις υπηρεσίε θα μπορούσε να αποτελέσει και πρότυπο για το πώς θα πρέπει να συζητώνται διαφορετικόμενα θέματα στο μέλλον. Η επόμενη λοιπόν ε, μεγάλη πρόταση ε, σε κάποιο θέμα ε, ίσως να γίνει έτσι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικρίνουν ε, εξυμνεί σε κάποιες περιπτώσεις το κοινοβούλιο. Είναι πάντα σοβαρό λοιπόν για το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει για να περάσει αυτή η πολύ σοβαρή νομοθεσία και η δουλειά του πραγματικά έφερε αποτελέσματα. Μπορεί να δημιουργήθηκε κάποια δυσαρέσκεια στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και... αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν είχαμε καμία άλλη ελπίδα να περάσουμε αυτή την πρόταση εάν δεν είχαμε ακολουθήσει αυτή την προσέγγιση και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πάντες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη βοήθειά τους. Η κυρία Γκέπχαρτ, ο Μάλκορ Χάρπορ, ε, τη συνεργασία από όλες τις πολιτικές ομάδες. Βάσει αυτής της συνεργασίας πέρασε η οδηγία για τις υπηρεσίες. Όχι η οδηγία που είχε ξεκινήσει το 2004, διότι αν είχαμε κάνει ακόμα εκείνη την πρόταση δεν θα είχε περάσει οδηγία για τις υπηρεσίες δεν θα είχαμε τίποτα σήμερα. Και ακόμα δηλώσεις θα κάναμε όλοι οι βαρύγδουπες και θα, ακούσαμε, θα ακούγαμε επικρίσεις ε, από όλες τις πλευρές. Δεν θα είχαμε οδηγία για τις υπηρεσίες. Το ερώτημα λοιπόν του Μάλκον Χάρπορ είναι το εξής. Η οδηγία για τις υπηρεσίες που έχουμε θα κάνει αυτό που θεωρήσαμε εμείς ότι θα έκανε η οδηγία για τις υπηρεσίες στη συμβιβαστική μορφή με την οποία πέρασε. Αυτό δεν θα το ξέρουμε ε, σύντομα. Πρέπει να περάσει κάποιο χρόνο. Πρέπει τα κράτη-μέλη να πάρουν το χρόνο του για να ολοκληρωθεί η διαδικασία εφαρμογή και μόνο στο μέλλον θα ξέρουμε τι θα γίνει. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι η οδηγία για τι υπηρεσίε, αν εφαρμοστεί με τον τρόπο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, θα δώσει μια πολύ σημαντική όθηση στι οικονομίε τη Ευρώπη. Το πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Ο Μάλκολ Χάρμπορ έθεσε μια ερώτηση σε αυτό το πλαίσιο ποια είναι η άποψή μου για το κατά πόσο όλα τα κράτη-μέλη πραγματικά θέλουν να έχουν μια πραγματική εσωτερική αγορά και έχει προχωρήσει περισσότερο το 2009 από το 1999. Αυτό ε, αφορά και άλλες πτυχές. Νομίζω ότι ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους αυτής της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης είναι ότι θα υπάρχουν κράτη-μέλη που δεν θα κοιτάνε προς τα έσω. Είναι φυσικό. Επειδή εγώ ήμουν πολιτικός αρκετά χρόνια, είναι φυσικό να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Όταν υπάρχει πίεση σε ένα κράτο μέλο, οι πολιτικοί πρέπει να αντιπακροθούν, το εκλογικό σώμα περιμένει να γίνει κάτι και ε, τις περισσότερες φορές κοιτάμε να δούμε τι μπορεί να γίνει εδώ και τώρα. Και αυτό είναι λογικό γιατί τα προβλήματα είναι εδώ και τώρα και προσπαθούμε να απαντήσουμε με αυτόν τον τρόπο και συχνά η πρόκληση είναι να χάνουμε την ευρύτερη εικόνα και να υιοθετούμε μέτρα τα οποία ε, θα αντιμετωπίσουν μερικώς το θέμα του εδώ και τώρα, αλλά μακροπρόθεσμα μπορεί να βλάψουν την όλη διαδικασία. Ε, νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα μεγάλα τεστ που πρέπει να ε, περάσουμε και να εφαρμόσουμε σε αυτή τη διαδικασία. Να μην εγκρίνουμε μέτρα μόνο για να αντιμετωπίσουμε το εδώ και τώρα που αργότερα θα έχουν μακροπρόθεσμες συνέπειες. Υπάρχουν ρώτησε ο κύριος ε, Χάρμπορ αν κάποια κράτη-μέλη απλά γλύφουν εντό εισαγωγικών ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις στις οποίες όντως συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αν συνεχίσουμε όμως να πιέζουμε και προσπαθήσουμε να κάνουμε τα θεμελιώδη βήματα, το κέρδος ε, συνολικά θα είναι καλύτερο από αυτό που θα χάσουμε ε, περιοδικά. Ε, ο κύριος Χάρμπορ αναφέρθηκε στο θέμα των κρατικών προμοθειών και το ανέφεραν και άλλοι συνάδελφοι. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις Αυτό παρεπιπτόντως επηρέασε και τις ε, συνθήκες και τις προϋποθέσεις που εφαρμόζουν κράτη-μέλη. Έχουν γίνει αρκετές μελέτες για το θέμα αυτό τα τελευταία χρόνια και τα κράτη-μέλη έχουν τη διακριτική ευχέρεια να κάνουν καταμερισμό μιας προμήθειας αν το επιθεμό. Παρά να έχουν ένα μεγάλο ε, μειοδετικό διαγωνισμό μπορούν να κάνουν μια κατανομή. Κάποια κράτη-μέλη δεν επιλέγουν να κάνουν κάτι τέτοιο. Ίσως μια νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να εξετάσει το θέμα και να δει τι θα γίνει. Ε, ίσως θα μπορούσαμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία των κρατικών προμηθειών και να δούμε ότι υπάρχουν και κάποιες αλλαγές. Το ανέφερα και αυτό, θα γίνουν και κάποιες αλλαγές το 2009-2010. Τα πιο νέα κράτη-μέλη, και τέθηκε και αυτό το ερώτημα στα πλαίσια αυτού του θέματος, εγώ ε, πιστεύω και στα νέα κράτη-μέλη και πιστεύω ειλικρινά ότι στα επόμενα 20 χρόνια άμα ανοίξουμε λίγο τα θέματα στις δημόσιες προμήθειες και κάνουμε πράγματα σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο για την εσωτερική οικονομία αλλά και για την όλη δημοκρατική διαδικασία αυτών των χωρών και αυτή είναι πραγματικά άποψη του Μαγκρίβη, δεν είναι άποψη του Επιτρόπου ότι σε 20-25 χρόνια όλα τα νέα κράτη-μέλη, κάποια ίσως καλύτερα από άλλα, αν όλοι λοιπόν έχουν διαφανείς ανοιχτές κρατικές προμήθειες, και γίνουν τα πράγματα με διάφανο τρόπο, σαφώς θα έχουμε όφελος για τις οικονομίες μας. Αλλά όλο αυτό δεν θα πρέπει να είναι ξεχωριστό από την όλη δημοκρατική και πολιτική διαδικασία. Αυτή είναι προσωπική μου άποψη, το επαναλαμβάνω. Τέθηκε επίσης κάποια ερώτηση για, τις, για τα διπλώματα ευρεσιτεχνία. Θα ήθελα πραγματικά να σας πω ότι τον Ιανουάριο του 2009 έχει διευθετηθεί το θέμα. Δυστυχώς δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Και η Γαλλική Προεδρία δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Προσπαθήσαμε να το παρακάμψουμε από διάφορες πλευρές. Είχαμε μικρή επιτυχία. Οι εσωτερικές υπηρεσίες μας κάναν τεράστια προσπάθεια για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία, αλλά εκεί που φαινόταν να λύνουμε ένα ε, λιθαράκι του προβλήματος, ξαφνικά ξεπηδούσε κάτι άλλο σε κάποιο άλλο τομέα. Πραγματικά λοιπόν δεν μπορώ να πω στον κύριο Μάντερς ότι το 2009 θα ολοκληρώθει αυτό το θέμα και θα τελειώσουμε στην Τσεχική Προεδρία. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο ρεαλιστές. Δεν μπορεί να τελειώσει το ζήτημα αυτό. Ο κύριος Μάντερς έθεσε επίσης το θέμα για το τι προκύπτει λόγω του ανταγωνισμού στις διαδικασίες επί παραβάση, το γεγονός ότι πρέπει να αποστέλλονται πίσω κάποια πράγματα. Ξέρω ότι αυτό το θέμα συζητήθηκε. Εξ όσων γνωρίζω, νομικός δεν είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο. είναι κάτι στο οποίο συμμετέχω αυτή τη στιγμή και ψάχνω να βρω και καλύτερε συμβουλές, αλλά προς το παρόν δεν μπορεί να γίνει. Κύριε Σφάμπ, σας ευχαριστώ πολύ για τη δουλειά σας. Συνεργάστηκα με πολύ χαρά μαζί σας. Ε, κάναμε πολύ καλή δουλειά στην Επιτροπή. Η ερώτησή σα ήταν κατά πόσο τα κράτη-μέλη είναι διατεθειμένα να συνεργαστούν καλύτερα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι θεωρείτε ότι έχει γίνει καλύτερα τώρα από ό,τι πριν από πέντε χρόνια. Δεν νομίζω ότι σε αυτή τη, ε, φάση μπορούμε να πούμε ότι όντω συμβαίνει αυτό. Ε, και αυτό είναι λόγω του οικονομικού κλίματο, όχι μόνο τη οικονομική κρίση στου τελευταίου μήνε. Το θέμα του Ιρλανδικού δημοψηφίματος αναφέρθηκε από κάποιους από τους ε, συναδέλφους. Νομίζω όμως ότι όλα τα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή, δεν έχω πάει σε κανένα από τα 27 κράτη-μέλη, όπου να βρέθηκε κάποιος και να μας είπε να δώσουμε περισσότερη εξουσία στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Από οποιαδήποτε πτυχή. Γνωρίσατε εσείς κανέναν από εσά να λέει κάτι τέτοιο. Αυτό που ακούγεται είναι ότι λογικά θα θέλαμε να τα κάνουμε μόνοι μας, ε, δεν θέλουμε να μας επιβάλλουν δικτατορικά την άποψή τους, δεν το θέλαμε αυτό κλπ. Εγώ μετά από πέντε χρόνια εδώ, ειλικρινά αυτή την ε, εκτίμηση κάνω. Η πολιτικοί κύκλοι και οι επιχειρηματικοί και οι οικονομικοί κύκλοι δεν είναι διατεθειμένοι να το κάνει αυτό και το ξέρω αυτό και αυτή την εκτίμηση, αυτή την εκτίμηση έχω καταλήξει ε, μετά από πέντε χρόνια εδώ. Έτσι έχει η κατάσταση. Βέβαια εμείς δεν μπορούμε να παραιτηθούμε διότι ούτως ή άλλως ε, πρέπει να πιέσουμε, πρέπει να κάνουμε διαπραγματεύσεις, πρέπει να γίνουν πολιτικές διαδικασίες για να προχωρήσει το θέμα αλλά δεν νομίζω ότι θα γίνει εύκολα υπάρχει και αυτή η ιδέα μιας συγκεκριμένης ημερομηνία. Έχει παρουσιαστεί αυτό το θέμα, αλλά δεν θέλουμε να καθορίσουμε ημερομηνία. Προσπαθήσαμε να συμφωνήσουμε σε αρκετούς τομείς. Υπάρχουν όμως δύσκολες αποφάσεις περί ανταγωνισμού που δεν μας επιτρέπουν να βρούμε περιθώριο να λειτουργήσουν τράπεζες και άλλα επιστοτικά ιδρύματα. Ελπίζω ότι η κρίσιμη μάζα θα μπορέσει να μετακινηθεί μέχρι το τέλος του έτους, διότι το Νοέμβριο του 2009 είναι περίοδος κλειδί για όλη αυτή τη διαδικασία και ελπίζω να έχουμε κάνει κάτι για αυτό το θέμα. Ο κύριος Βάμπε έθεσε και κάποιο θέμα για τις προμήθειες και την ευελιξία. Οι κανόνες μας ε, αφήνουν αρκετό περιθώριο ευελιξία σε κράτη-μέλη. Ίσως σε κάποιους τομείς θα μπορούσατε να πείτε ότι η ευελιξία είναι κάτι που δεν θα έπρεπε να έχουν, αλλά, ε, γιατί θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με λανθασμένο τρόπο, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε στο μέλλον. τέθηκε και το θέμα των τηλεπολίσεων και τη χρήση των πιστοτικών ε, καρτών και κάποιους περιορισμούς. Ναι, γνωρίζω ότι υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Ε, έχω και κάποια προσωπική πείρα επί του θέματος και αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα, το γεγονό ότι δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει κάποιο την πιστοτική του κάρτα, είναι κάτι το οποίο πρέπει να εξετάσουμε και να δούμε τι μπορεί να γίνει. Νομίζω ότι αυτό όντω αποτελεί περιορισμό τη ελεύθερη αγορά. Δεν ξέρω όμω νομικά τι γίνεται για το θέμα αυτό, αν είμαστε εντό ή εκτό κανόνων, αλλά είναι κάτι το οποίο προέκυψε πρόσφατα και έχουμε λίγη πείρα με το θέμα. Ο κύριος Χάσε Φερέρα αναφέρθηκε πολύ εύγλωτα στην μεταφορά τη οδηγία για τις υπηρεσίες. Δεν θέλουμε να κατονομάσουμε κανέναν. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποιο θα έχει πάει καλά και κάποιο όχι. Το θέμα της μεταφοράς είναι κάτι το οποίο προχωράει σε αρκετά κράτη-μέλη. Ε, θα δούμε τι θα γίνει και στο, μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε μια αξιολόγηση. Εγώ επαναλαμβάνω σε όλα τα κράτη-μέλη να υπάρχει αρκετό προσωπικό να έχουν πόρου ε, προσωπικό για την εφαρμογή τη οδηγία για τι υπηρεσίε. Κάποιο υπουργό από ένα κράτο μέλο ήρθε πριν από ένα χρόνια και Συζητώντα το θέμα τη εφαρμογή μου είπε ότι θα χρειαστούν τεράστια δουλειά όλες οι διοικητικέ υπηρεσίες για να μπορέσουν να εφαρμόσουν οδηγία για τι υπηρεσίες. Και Ακόμα και από τη χώρα που ξέρω καλύτερα όντως ε, το ίδιο πράγμα μου λένε. Όντως θα καθυστερήσει το θέμα. Δεν νομίζω ότι η νομική κρίση θα επηρεάσει την εφαρμογή της ε, οδηγίας για τις υπηρεσίες. Ακόμα και αν λόγω της κρίσης κάποια κράτη-μέλη κοιτάνε πιο πολύ τα εσωτερικά τους θέματα και όχι τα ευρωπαϊκά. Ο Πρωθυπουργός μου, από ό,τι γνωρίζω εγώ στην Ιρλανδία, έχει δεσμευτεί να το θέσει το θέμα αυτό στους Ιρλανδούς ε, ξανά και να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Ε, το τι μπορεί να συμβεί τον Ιανουάριο ή τον Μάιο μπορεί να είναι διαφορετικό τον Ιανουάριο του 2009 μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που θα γίνει το φθινόπωρο του 2009 ε, αυτό λέει και η πολιτική μου πείρα ε, έγινε μια εκστρατεία για, την, ε, για το προηγούμενο δημοψήφισμα και πιστεύω ότι οι Ιρλανδοί τελικά θα μπορέσουν να, το, να καταλήξουν σε μια απόφαση. Η κυρία Πλεστίνσκα, την ξέρω πάρα πολύ καλά από τη Σλοβακία, για το One Stop Stop, αυτή τη μία και μόνη θηρίδα. Ε, θα κάνουμε μελέτες για να δούμε τι συμβαίνει, πού έχουμε καλά αποτελέσματα, αλλά δεν μπορούμε να αρχίσουμε να το κάνουμε αυτό πριν το 2010, όπου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Δεν ξέρω αν θα χρησιμοποιήσουμε το benchmarking, αλλά πάντα μαθαίνουμε από τις βέλτιστες ε, πρακτικές και θέλουμε να δούμε τι θα γίνει με το θέμα αυτό. Για το θέμα του γεγονότος ότι δεν επωφελούνται πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τις δημόσιες ε, προμήθειες, ε, ίσως θα έπρεπε να ξαναδούμε λίγο τους κανόνες διότι άκουσα από πολλούς ε, το θέμα για τις δημόσιες προμήθειες. Ίσως ο νέος επίτροπος λοιπόν θα μπορούσε να το εξετάσει το θέμα. Η κυρία Βάιλερ ε, αναφέρθηκε στο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέματα που σχετίζονται με αυτό. Εγώ είμαι αισιόδοξο. Εμένα δεν με νοιάζει να κάνουμε τρία βήματα μπροστά και δύο πίσω. Πάλι έχουμε κερδίσει ένα βήμα. Αυτό λοιπόν έχει σημασία, να συνεχίσουμε να προχωράμε μπροστά. Αυτό που θέλω να κάνω πάντα είναι να είμαι ρεαλιστής και πρακτικός για τα θέματα αυτά. Τώρα, για το θέμα το... της συνεργασίας με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Όντως έχουμε πολύ ψηλό επίπεδο συνεργασίας με τις Ηνωμένε Πολιτείες συνδιαλεγόμεθα. Αυτά ε, τα βρήκα ούτως ή άλλως έτοιμα εγώ πριν έρθω. Ήταν θεσπισμένα τα πάντα. Δεν μπορούμε πάντα να συμφωνούμε σε όλα, αλλά και οι δύο πλευρές ε, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει από την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Σε κάποιους άλλους τομείς ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα, αλλά η ιδέα ενός διατλαντικού οικονομικού συμβουλίου και οι συζητήσεις ε, με την Αμερική ξεκίνησαν το 2007, ξεκινήσαμε, είχαμε πολλά, πολύ καλά αποτελέσματα, κάναμε μια επόμενη συνεδρία στο Δεκέμβριο και ελπίζομαι η νέα κυβέρνηση Ομπάμα να ε, συμμετέχει τόσο ενεργά και να είναι τόσο δεσμευμένη όσο η προηγούμενη κυβέρνηση. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να συζητήσουμε και όχι μόνο τους δημοσιονομικούς κανονισμούς. Χαίρομαι ιδιαίτερα για τα σχόλια της Σάρλοτ όπως και οι περισσότεροι, ξέρει πολύ καλά πώς δουλεύω. Προσθέτω και ένα ψύχμα ρεαλισμού σε όσα κάνω. Και ελπίζω για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 25 χρόνια να υπάρχουν άνθρωποι που να πούνε ότι όντως προχωρήσαμε. Μετά από τα δύσκολα οικονομικά προβλήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση προόδευσε και καταφέρνει να κάνει τα πράγματα στα οποία είμαστε καλοί. Εγώ πραγματικά ε, βασίζω τις ελπίδες μου σε αυτό. Κυρία Πρόεδρε, θέσετε το θέμα του ρόλου των νέων κρατών μελών. Δεν το λέω γιατί είστε εσείς πρόεδρος εδώ, το έχω πει και σε άλλες ε, περιπτώσεις δημοσίως. τα, εσείς ως κρατημέλη είστε πιο δεσμευμένοι στο άνοιγμα της αγοράς από τις παλιότερες χώρες. Ε, είχαμε πάρα πολύ καλές θετικές, πολύ θετικές εκθέσεις και ελπίζω αυτό να συνεχιστεί και ελπίζω η επιρροή τους να ε, περάσει και στα παλιότερα κράτη-μέλη και να περάσουμε σε μία περίοδο που θα έχουμε καλύτερες αξιολογήσεις. Τα νέα κράτη-μέλη είναι πάρα πολύ ανοιχτά στην ιδέα της εσωτερικής αγοράς, ε, διαπιστώνουν ότι όντως υπάρχουν ευκαιρίες και προσπαθούν να τις αναζητήσουν. Ευχαριστώ πολύ για τα λόγια σας, για τη δουλειά σας, για τη συνεργασία μας. τα τελευταία πέντε χρόνια. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους για τις ερωτήσεις που έθεσαν, για τις παρατηρήσεις που έκαναν. Θα ήθελα να κλείσουμε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη. Και ελπίζουμε να σας δούμε κάποια στιγμή ε, να πιούμε ένα ποτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, μην φύγετε. Έχουμε τίποτα στα διάφορα. Όχι. Απομένει η ημερομηνία της επόμενης συνεδρίασης. Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου. Και την επόμενη Τετάρτη και Πέμπτη, 11 και 12. Ε, καλό Σαββατοκύριακο.